Diamo inizio colleghi. Possiamo riprendere. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε από το σημείο 9. Το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Πολύ γρήγορα συνάδελφοι γιατί έχουμε και ψηφοφορία γεωργικές στατιστικές της αλίας. Πρόκειται για ένα κείμενο ευθυγράμμισης με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ας περάσουμε στην ψηφοφορία στο σχέδιο της Επιτροπής, σχέδιο κανονισμού που τροποποιεί ορισμένες νομοθετικές πράξεις στον τομέα των γεωργικών και αλλιευτικών στατιστικών. Ως ε, ε, εισηγητής. Θεωρώ ότι η πρόταση ευθυγράμμισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως έχει δεν μας παρουσιάζει προβλήματα. Έχω συμπεριλάβει μόνο εννέα ταυτόσιμες ε, τροπολογίες, μία για κάθε τροποποιητική πράξη σύμφωνα με τους κανόνες της θεσμικής συμφωνίας μεταξύ των τριών οργάνων για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Ε, για, την περίοδο της εξουσιοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η περίοδος ε, για να εκδώσει τις κατεξουσιοδότηση πράξης δεν πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας, αλλά πρέπει να περιορίζεται σε μία πενταετία. Δεν υπάρχουν άλλες τροπολογίες από τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας Ωστόσο, στο μεταξύ ενημερωθήκαμε ότι το Συμβούλιο προτείνει καινούργιες τροπολογίες, οι οποίες είναι προβληματικές για τις θέσεις του Κοινοβολίου. Για θέματα ευθυγράμμισης, όπω τα συζητήσαμε και χθε. εάν το Συμβούλιο επιμείνει στις θέσεις του, θα πρέπει να οργανωθεί ένας τριμερός διάλογος. Διαφορετικά μπορούμε να προχωρήσουμε με τη δική μας θέση. Συνάδελφοι, αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις και αιτήσει παρέμβασης, προτείνω να ψηφίσουμε και αν συμφωνείτε να, να ψηφίσουμε συνολικά. Εάν συμφωνείτε λοιπόν και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, ηλεκτρονικά. Α, ναι. Απαιτείται η τελική ψηφοφορία να είναι ηλεκτρονική. Επομένως βγάλτε τις κάρτες. Αν είστε όλοι έτοιμοι λοιπόν, κυρίσω την ψηφοφορία. Θέτω σε ψηφοφορία όλες τις τροπολογίες μαζί. Υπέρ. Ψηφίστε. Αν κάποιος δεν έχει την κάρτα, να το πει, για να το σημειώσει η γραμματεία. Εντάξει, ωραία, υπάρχει ομοφωνία. Ευχαριστώ. Και τώρα, τελική ψηφοφορία για, την, ε, για το σχέδιο όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ε, τώρα άνοιξε η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα... Ας προχωρήσουμε συνάδελφοι. Σημείο 10. Παρουσίαση από την Επιτροπή της νομοθετικής πρότασης σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις για το 2014. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι μεταβατικές διατάξεις το 2014 πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι το τέλος του έτους. Ως μεταβατικές διατάξεις είναι οι τεχνικές ε, διατάξεις για την συνέχεια των διαφόρων μορφών στήριξης στήριξης της γεωργικής πολιτικής για το 2014. Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να αναλάβουν νομικές υποχρεώσεις για οποιοδήποτε μέτρο στο πλαίσιο της, αγροτικής της ανάπτυξης της υπαίθρου που ήδη έχουν εγκριθεί το 2014 με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να είναι επιλέξιμες και για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Ε, οι μεταβατικές λοιπόν διατάξεις περιλαμβάνουν και το νέο κράτος μέλος, στην Κροατία και επιτρέπουν στα εθνικά κοινοβούλια να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το 2014 τα ισχύοντα. Εξάλλου, χθες αποφασίσαμε στην συνάντηση των, στη συνεδρίαση των συντονιστών το ΕΛΚ να αναλάβει αυτήν την ευθύνη να, να, να είναι οι εισηγητές δηλαδή. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Χανιώτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να μας παρουσιάσει την πρόταση και ζητώ από τους συναδέλφους να εγγραφούν στη λίστα των αγορητών. Κύριε Χανιώτη, έχετε το λόγο. Oh, uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τα μέλη της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής που μου δίνουν την ευκαιρία να κάνω μια σύντομη εισαγωγή όσον αφορά την προσέγγιση από πλευράς uh, ε, διάρθρωσης αυτής της πρότασης. Τώρα, εδώ σε σχέση με τα θεσμικά όργανα μέσα στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων για την προαγωγή της μεταρρύθμισης της ε, αγροτικής πολιτικής και την προσπάθεια να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014 πρέπει να πούμε ότι τούτου λεχθέντος υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία από πλευράς νομικής βάσης ε, που σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου προβλέπονται κάποιοι μεταβατικοί κανόνες που θα χρειαζόμαστε Merci. για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια χωρίς προβλήματα μετάβαση σε αυτό το νέο σύστημα και θα διασφαλιστεί και η συνέχεια και συνεκτικότητα. Αυτή είναι η λογική που εμπνέει αυτή την προσέγγιση από πλευρά μα. Όσον αφορά τι άμεσε πληρωμέ, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες πληρωμών των κρατών μελών να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο για αυτή την έναρξη αυτού του νέου συστήματος. Πράγμα το οποίο θα απαιτήσει κάποιες προσαρμογές για τον τρόπο με τον οποίο θα χορηγείται η βοήθεια. Επίσης θέλουμε να επιτρέψουμε να έχουν χρόνο οι γεωργοί να πληροφορηθούν για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η νέα πολιτική. Γι' αυτό τα αιτήματα για το 2014 θα εξεταστούν υπό αυτούς τους προσωρινούς κανόνες που θα λαμβάνουν επίσης υπόψη και την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το δεύτερο πυλώνα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να μπορέσουμε δύο αλληλοδιάδοχες περιόδους να τις ε, ε, καταστήσουμε συνεκτικές ε, με ειδικά μέτρα. Είναι κάποια νέα στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη που απαιτούν εξειδικευμένες τέτοιες ε, διατάξεις και ρυθμίσεις. Πρώτα απ' όλα, η καθυστέρηση της απόφασης ε, για τις νέες άμεσες πληρωμές συνεπάγεται ότι πρέπει κάποια θέματα να αποσαφινιστούν όσον αφορά τη βασική γραμμή που θα ισχύει όσον αφορά τα μέτρα τα αγροπεριβαλλοντικά στον τομέα της γεωργίας και την εφαρμογή της διασταυρούμενης συμμόρφωσης, της πολλαπλής συμμόρφωσης. Υπάρχει επίσης η ανάγκη για κάποιες ε, μεταβατικές ε, διατάξεις και ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να αναλαμβάνουν ε, υποχρεώσεις όσον αφορά την εκτινοτροφία για το 2014 ακόμα και αν έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια για την τρέχουσα περίοδο και δίνοντας τη δυνατότητα να συνεχίσουν οι δεσμεύσεις μας όσον αφορά την, ε, το πλαίσιο της νέας δημοσιονομικής περίοδου. Και τέλος, για τον οριζόντιο κανονισμό υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν κάποια μεταβατικά μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν, για παράδειγμα, να συνεχιστεί το πρόγραμμα ΑΙΑΚΑ και το σύστημα της πολλαπλούς συμμόρφωσης ε, σε σχέση με τις απαιτήσει του νέου συστήματος. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ το γεγονός ότι τα προσωρινά μεταβατικά μέτρα συμπεριλαμβάνουν διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ πυλώνων για τα κράτη-μέλη, παρένθεση ελαστικότητα και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το MFF. Σε αυτό το πλαίσιο της ελαστικότητας για τη μεταφορά κονδυλίων μεταξύ πυλώνων, το γνωρίζουμε καλά και το έχουμε σημειώσει ότι και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν υιοθετήσει θέσεις που πρέπει να οδηγήσουν σε κάποια προσέγγιση και συμφωνία. Γι' αυτό όλες οι αναφορές που κάναμε στο IMFF αναφέρονται σε παρένθεση ώστε να επιτρέψουμε να υιοθετηθεί ο κανονισμός με την ε, λήψη τελικής απόφασης από πλευρά τους για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η μείωση άμεσων πληρωμών είναι κατ' εκτίμηση 130 εκατομμύρια για την περίοδο 2015 που αφορά τις ε, αιτήσει ε, για το 2014 για τις άμεσες πληρωμές και σε σχέση με τα μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου θα υπάρξουν κάποιες μεταφορές αλλά χωρίς σημαντική οικονομική επίπτωση συνολικά. Δεν μπορούμε να ποσοστοποιήσουμε αυτή τη στιγμή σε ακριβή μεγέθη αυτά τα ποσά. Αυτά είναι γενικά αυτά τα οποία βρίσκονται και καλύπτουν το, τους στόχους αυτής της μεταβατικής ρύθμισης. Ε, και είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις να απαντήσω και να διευκρινίσω αν απαιτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Molto Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, Τάσο. Νομίζω ότι τα παρουσίασες πολύ ωραία. Ντόρφμαν. Θεία Πέρες, παρακαλώ, η Ράτσα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ απλά ζήτησα τον λόγο για να διατυπώσω κάποια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, να ευχαριστήσω για την παρουσίαση βέβαια. Έχω την εντύπωση όμως ότι επαναλαμβάνουμε κάπως τα ίδια επιχειρήματα όπως και χθες σε σχέση με τον κανονισμό δημοσιονομικής πειθαρχία. Αυτός ο κανονισμός πρέπει να γίνει φυσικά, διότι πρέπει να έχουμε ένα μέσο στα χέρια μας για να απαντήσουμε και να αντιδράσουμε σε σχέση με τα αιτήματα των γεωργών για το επόμενο έτος, μια και δεν μπορεί να αρχίσει άμεσα έτσι να εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση. Αλλά επίσης και αυτός ο κανονισμός έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών έτσι λοιπόν βλέπω κάποια αριθμητικά μεγέθη, κάποια ποσά, κάποιες τροποποιήσεις που υπάρχουν όσον αφορά τα παραρτήματα. Ένα σε σχέση με το παράτημα 8, σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις ανακράτος. Και θεωρώ ότι έγιναν κάποιοι υπολογισμοί με βάση αυτή τη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το Ευρωκοινοβούλιο, η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ζητούμε να μας δοθούν τα στοιχεία ανακράτο. Μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή της. Είναι το Συμβούλιο λέει που έλαβε αυτή την απόφαση. Αλλά αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη αυτού του παρατήματος. Και ερώτηση. Αυτές οι μειώσεις που εξετάζονται είναι επίπτωση της εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας ή μήπως είναι σε σχέση με την ε, ε, ε, αυξημένη εφαρμογή, αύξηση της εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είναι θέμα υπολογισμών βέβαια και μπορώ να υπολογίσω το τι συμβαίνει. Επιμένω και μένω όταν λέει ο Υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας ότι εμείς θα έχουμε περισσότερα λέει κονδύλια για την ΚΑΠ για την επόμενη περίοδο, βλέπω εδώ στο παράρτημα ότι για την περίπτωση της Ισπανίας, της χώρας μου ακριβώς, υπάρχει μια μείωση γύρω από το 6,25% μείωση. Από 5.150.000 πάμε στα 4 τόσα εκατομμύρια. Μπορεί να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό είναι εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο παραπάνω να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται σε βάση με αυτά τα οποία έγιναν οι υπολογισμοί και συντάχθηκε αυτό το παράρτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Herbert και μετά το λόγο πάει στον Κώστα. Ο κύριο Ντόρφμαν, ευχαριστώ θερμά πρόεδρε. Η πρώτη μου ερώτηση προ την ίδια κατεύθυνση στοχεύει, όπω η ερώτηση τη συναδέλφου Ιράτσε, που ήθελε απλά και μόνο μία επερώτηση να διατυπώσει διαδικαστικά. Αυτή τη μεταβατική περίοδο η αντιμετώπιση πρέπει να την εξετάσουμε στο Κοινοβούλιο. Όπως μας είπε ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται και είναι αυτονόητο αυτό για οικονομικούς κανονισμούς και υπολογισμούς. Το κάνουμε αυτό ούτως ή άλλως για τον προϋπολογισμό για του χρόνου. Δεν θα υπάρχουν πολιετής προϋπολογισμοί. Πώς αυτά τα δύο θα συνδεθούν μεταξύ τους. Αυτές οι μεταβατικές προσωρινές ρυθμίσεις μπορούν να εγκριθούν προτού υπάρξει καν συνολικός προϋπολογισμός. Δεύτερη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου τι κάνει Πώς έχει το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη ή οι περιφέρειες, τα κρατήδια ή πρέπει να υποβάλουν τα σχέδια για την ανάπτυξη της υπαίθρου όπως το 2013 ή θα είναι μεταβατικές ρυθμίσεις για το 2014 περισσότερο που τα κράτη-μέλη θα καταρτίζουν αυτά τα προγράμματα και τα σχέδια αυτά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μέχρι τα τέλη αυτού του έτους σε ένα κράτος μέλος και σε όλες τις περιφέρειες, παράδειγμα έχω υπόψη μου τη Γερμανία, ε, την Ιταλία όπου υπάρχουν πολλά προγράμματα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλα αυτά για την ανάπτυξη Συπέθρου την 31η ε, ε, Δεκεμβρίου 2013 θα έχουν εγκριθεί και έτσι αμέσως θα έχουν έχουν υποβληθεί και θα εγκριθούν αμέσω από την Επιτροπή μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χέρπετε. Λουίς Καπούλα Σάντος. Ναι, ε, μετά ο τάσο. Ο Λουίς, ο Λουίς μετά ο Τάσος. Το κυριότερο τμήμα τη ερώτηση που ήθελα να θέσω πολύ καλά διατυπώθηκε από τη συνάδελφο Ιράτσε διαπιστώνω ότι υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ. Πρώτον, εμείς ακόμα δεν έχουμε συζητήσει ούτε στον τριμερή διάλογο το θέμα της εξωτερικής σύγκλησης. Και εδώ έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρεί δεδομένη την κατάσταση σε σχέση με την πρόταση του Συμβουλίου. Θεσμικά λοιπόν πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη ευγένεια εναντί του Ευρωκοινοβουλίου κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν να μην υπάρχει το Κοινοβούλιο, σαν να είναι ανύπαρκτο το Ευρωκοινοβούλιο και αυτό είναι κάτι απόλυτα παράδεκτο. Δεύτερη ερώτηση, περισσότερο πρακτικού χαρακτήρα που θέλω να διατυπώσω αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Από ό,τι είδα, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνάψουν νέες υποχρεώσεις στα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου μέσα στο 2014. Αυτό δηλαδή σημαίνει με άλλα λόγια το 2014 για την ανάπτυξη της υπαίθρου ακόμα θα είναι ένα έτος ανάληψης υποχρεώσεων και δεσμεύσεων. Ε, θα πρέπει αυτό να το δούμε για τα επόμενα δύο χρόνια και θα ήθελα να επιβεβαιωθεί, να επαλήθευθεί, αν πράγματι αυτό συμβαίνει στην πρακτική, πράγμα που σημαίνει ότι την έγκριση υποψηφιωτήτων σχεδίων και προγραμμάτων το 2014 θα είναι ίδιο έτος όπως οποιοδήποτε άλλο έτος για την λειτουργία αυτού του προγράμματος. Ήθελα απλά και μόνο αυτή την επιβεβαίωση, επαλήθευση αυτής της κατάστασης. Ευχαριστώ. Πριν δώσω τον λόγο στον Τάσο, θα ήθελα ωστόσο να κάνω μια διευκρίνηση μετά την παρέμβαση ε, του Λουίς Κάποντα Σάντος. Η έκθεση αυτή για τις μεταβατικές διατάξεις είναι μια νομοθετική πράξη όπως και κάθε άλλη. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι υπάρχει η ίδια ακριβώ διαδικασία συναπόφασης όπως και στους άλλους φακέλους της κοινή γεωργικής ε, ε, πολιτικής και συνδέεται στενά με τους τέσσερις άλλους φακέλους. Χθε στη συνεδρίαση των συντονιστών θέλησαμε να διευκρινίσουμε τη σημασία της συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης που συνδέεται πολύ στενά με τις άλλες. Και είναι σημαντικό να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ του εισηγητή αυτής της έκθεσης με τους εισηγητές των άλλων τεσσάρων φακέλων. Ακριβώς λοιπόν επειδή θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει πλήρης αρμονία μεταξύ των, αποφάσεων που θα ληφθούν στο πλαίσιο των άλλων τεσσάρων νομοθετικών πράξεων με, τα, με τις μεταβατικές διατάξεις ε, τις οποίες θα αποφασίσουμε για τη συγκεκριμένη νομοθετική πράξη. Να μην υπάρχει λοιπόν αμφιβολία εναντί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου ότι αυτή η νομοθετική πράξη συνδέεται στενά με τις άλλε και ότι το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το βλέπει αυτό υπό μια ενιαία λογική. Ο τάσο Χανιώτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγείρατε πολύ ορθά ζητήματα. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Κάπουλος Άντος. όχι μόνο σας σεβόμαστε ως όργανο και θεσμό, όπως το ξέρετε πολύ καλά, αλλά σας θεωρούμε και ένα όργανο, ένα θεσμό που θα παίξει κρίσιμο ρόλο στη συζήτηση και ε, ε, ε, πραγματικά αυτό ακριβώς έχει να κάνει με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον μη παραγωνισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φυσικά. Υπάρχει βέβαια ένα χρονοδιάγραμμα. Την 1η Ιανουαρίου του 2014, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα πρέπει να εγγυηθούμε μια ομαλή μετάβαση από το σημερινό σύστημα στο καινούριο σύστημα. Και για το λόγο αυτό ε, ο κανονισμός αυτός προσπαθεί να εντοπίσει ακριβώς τους τομείς εκείνους και στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου χρειάζονται τέτοιες μεταβατικές διατάξεις. Προφανώς, πώς θα γίνει η μετάβαση των άμεσων ενισχύσεων χωρίς να διευκρινιστούν τα ποσά, οι αριθμοί, αυτό δεν είναι δυνατόν. Ελπίζουμε και νομίζω όλοι εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση να έχουμε τους αριθμούς και τα ποσά, να τα διευκρινίσουμε το συντομότερο δυνατόν, γιατί διαφορετικά η μετάβαση θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε για την ανάγκη να έχετε τους ακριβείς αριθμούς και θα περάσω το μήνυμα αυτό και στους συναδέλφους που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι γνωρίζετε κι εσείς πώς έχει η κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου είναι ευκολότερο να βγάλουμε τα ποσά στις άμεσες ενισχύσεις, γιατί οι άμεσες ενισχύσεις αποφασίζονται κατά τρόπο που είναι διαφανής. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη σαφήνεια όσο αφορά τα θέματα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Εσείς ξεκαθαρίσατε τη θέση, τη θέση σας. Το έχουμε συζητήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Σέβομαι πλήρως τη θέση σας. Το τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να επισημάνω έχει να κάνει με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τα σχετικά μέτρα θα διακρίνονται από μια συνέχεια, αλλά θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές. Το πλεονέκτημα στην ανάπτυξη της υπαίθρου σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις είναι ότι υπάρχει μια ευελιξία στην κατανομή των πόρων στα διάφορα έτη. Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται πυρετιβώς για να, ε, και όλα τα κράτη-μέλη εργάζονται πυρετοδός για, να, για τα μελλοντικά τους σχέδια σχετικά με την ανάπτυξη της υπαίθρου και γίνεται και δουλειά για να διευκρινιστούν σε γενικές γραμμές οι στόχοι του προγράμματος αυτούς εντός του καλοκαιριού. Όταν θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες ε, αυτού, των πραγμάτων που θα συμφωνηθούν, θα μπορέσουμε να είμαστε πιο σαφείς. Υπάρχει επίσης το λεγόμενο greening, η, περιβαλλοντική ανάπτυξη, η ανάπτυξη με περιβαλλοντική συνιστόσα. Και αυτό θα είναι πολύ καθοριστική και θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο τα αγροδιατροφικά προγράμματα θα περάσουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Για άλλη μια φορά λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να εντοπίσουμε εδώ είναι να δούμε ποιοι είναι οι τομείς και τα μέτρα ε, με τα οποία θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μια ομαλή μετάβαση από τους υφιστάμενους κανόνες, αλλά να αφήνουμε και ένα περιθώριο για αναπροσαρμογές όταν διευκρινιστούν και όλα τα υπόλοιπα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν περιγράφω ποια είναι η λογική και τονίζω για άλλη μια φορά το γεγονός ότι τα πάντα συνδέονται με το πολιετές ε, δημοσιονομικό ε, πλαίσιο και υπάρχει πλήρης αναγνώριση και σεβασμός του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την επεξεργασία και οριστικοποίηση της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Τάσο. Ωραία. Νομίζω ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες διευκρινήσεις ε, πλέον. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να λάβουν το χολόγο. Όχι. Α, η Ράτσα, άλλη μια ερώτηση. Λυπούμε, αλλά σε σχέση με την αποσαφήνιση της αμφιβολίας που είχα πρέπει να πω ότι το 6,25% λιγότερα που φαίνεται από το παράρτημα της Ισπανίας είναι η εφαρμογή δημοσιονομικής ε, πειθαρχία ή είναι άλλες ε, μεγαλύτερες περικοπές. Πρέπει να το ξέρω αυτό γιατί είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο. Ε, τάσος. Ναι, Τάσο μπορείς να κάνεις άλλη μια διευκρίνηση. Αν και νομίζω ότι η απάντηση είναι θετική. Τάσο. Ναι, η απάντηση είναι καταφατική, αλλά θα προσπαθήσω να στείλω και πιο αναλυτικούς ε, πίνακες, έτσι ώστε η εικόνα να καταστεί σαφής. Ευχαριστώ. Sí. Ε, Πρόεδρος, ευχαρι... ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή και τον Διευθυντή Τάσο Χανιώτη. Η Ράτσε, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται ε, με την λογική της μεταφοράς ε, των αποτελεσμάτων της 8ης Φεβρουαρίου. Ε, σε αυτή τη λογική κινούμεθα, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και όπως είπε και ο συντονιστής Βίσκας, αλλά έχει ζητήσει και το ρόλο, το λόγο. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω με εκτίμηση προς τον κύριο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει αναγνωρίσει ότι τα μεγέθη για τον πρώτο πυλώνα υπολογίστηκαν με μεγαλύτερη διαφάνεια από ότι τα ποσά για το δεύτερο πυλώνα. Και υπογραμμίζω αυτό υπολογίστηκαν με μεγάλη. Ακόμα και όλα τα στοιχεία τα άλλα και του δεύτερου πυλώνα πρέπει με τη μέγιστη διαφάνεια να συντάσσονται και θέλουμε να διαβιβαστούν εφόσον πρέπει να γνωρίζουμε επίσης το πλαίσιο των δημοσιονομικών αυτών χαρτοφυλακίων για το τι αποφασίστηκε δηλαδή στο Συμβούλιο της 8 Φεβρουαρίου. Μια και προφανώς υπάρχει η διαπραγμάτευση που έχει κλείσει, μια και όλοι οι υπουργοί είπαν ότι σε σχέση με το Συμβούλιο ποια θα είναι τα ποσά τα οποία θα κατανέμονται στο δεύτερο πυλώνα για κάθε χώρα. Και φυσικά το Ευρωκοινοβούλιο, γι' αυτό το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερωθεί, μια και εμπλέκεται και έχει κάτι να πει για αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Θέλω να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, την παρουσίαση της μελέτης και του περιβαλλοντικού ρόλου των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην νέα κοινή γεωργική πολιτική χωρίς χρονοτριβές. Να ευχηθώ ε, το καλωσόρισες ε, στην ε, καθηγήτρια Κριστίνα Ρόρετς, η οποία θα μας παρουσιάσει μια έρευνα, μια μελέτη πάνω στα περιβαλλοντικά ωφέλη της ε, αύξησης της καλλιέργειας των πρωτεϊνούχων φυτών στο πλαίσιο της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής. Επίσης, ε, ευχόμαστε το καλωσόρισες και στους άλλους πέντε μελετητές, Πίτερ Ζάντερ, Ανδρέα Μπούς, Σάρα Πρέσελ, το Γερμανικό Φορέα για την Μελέτη του Περιβάλλοντος, τον Ντόναλτ Μάρφι Μπόρκαντ, Ντάρφι Πόρσκετ από τη Γερμανία. Δίνω αμέσω το λόγο στην δόκτωρα Βότσον για την παρουσίαση της μελέτης και ζητώ από τους συνεδέλφους να ζητήσουν να εγγραφούν στον κατάλογο των παρεμβάσεων. Κυρία Βότσον, 20 λεπτά. 20 λεπτά έχετε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτή τη μελέτη. Έχετε μπροστά σας ένα σχέδιο το σχέδιο της μελέτης. Από τότε που γράφτηκε όμως ήδη άλλαξαν τα πράγματα. Βασιζόμαστε στα επιστημονικά δεδομένα και σε εμπειρογνωμοσύνη με βάση των οποίων κάναμε τις συστάσεις μας αλλά και εσείς μπορείτε να κάνετε συστάσεις στην τελική μορφή των συμπερασμάτων. Αρχίζω υπενθυμίζοντας τι είναι τα οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Όλες ανήκουν στα λαχανικά στα όσπρια μάλλον, μεταξύ των οποίων και η Σόγια και ο Αρακάς χορηγούν αμινοξέα για την ανάπτυξη του οργανισμού. Το βασικό στοιχείο είναι ότι τα όσπρια κάνουν κάτι μοναδικό που είναι η, η χρήση του αζότου που είναι τελείως ιδιαίτερη στα όσπρια. Θα βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες ότι φαίνονται μερικοί κόκκι που είναι άζωτο το οποίο μαζεύουν από την ατμόσφαιρα. Επίσης έχουν ιδιαίτερο τρόπο άνθησης που το αναγνωρίζουν εύκολα οι κυπουροί. Όλοι γνωρίζουμε τα μπιζέλια και τα φασόλια και τα λούπινα και τις φακές, όλοι τις γνωρίζουμε. Άλλο σημαντικό στη, στοιχείο των οσπρίων είναι οι ζωοτροφές που χρησιμοποιούμε στα ζώα, το τριφύλι, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες έχω στην ε, προσθήκη. Στην προσθήκη. η κτηνοτροφία στην Ευρώπη εξαρτάται από εισαγόμενες πρωτεΐνες. Δέστε τους αριθμούς εδώ τη γραφική παράσταση στα αριστερά. Βλέπετε ότι συνεχώς αυξάνονται οι εισαγωγές πρωτεϊνούχων όπως τη σόγιας. Και επίσης εκεί δείχνουμε και τις τιμές, την εξέλιξη των τιμών με την διακεκομένη και τη συνεχή γραμμή συνεχώς αυξάνεται και η τιμή. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις για τις μελλοντικές μας εισαγωγές. Μπορούμε να τα σκεφτούμε ως ποσότητες μεν, αλλά μπορούμε να το αναλύσουμε σύμφωνα και με το πώς η γη καλλιεργείται για αυτά τα πρωτεϊνούχα. Στο στη δεξιά γραφική παράσταση λοιπόν δείχνουμε ότι υπάρχουν εξαγωγές υδατανθράκων αλλά εισαγωγές πρωτεϊνών. 15 εκατομμύρια εκτάρια περίπου χρησιμοποιούνται. Σήμερα το ποσοστό γεών που χρησιμοποιείται για πρωτεϊνούχα στην Ευρώπη είναι χαμηλό. Ακόμη και τα σκοτεινότερα σημεία εδώ στο χάρτη δείχνουν μόνο 8 με 25% να χρησιμοποιείται για πρωτεϊνούχα και τα υπόλοιπα τα σκιασμένα είναι πολύ λιγότερη γη. Τώρα για ένα γεωργό που παράγει πρωτεϊνούχα το κύριο όφελος είναι ότι χρειάζονται λιγότερα λιπάσματα, ζωτούχα λιπάσματα γιατί είναι πιο οικονομική η χρήση τους χρησιμοποιείται και για την επόμενη καλλιέργεια. Δηλαδή δεύτερο όφελος. Η εναλλαγή των καλλιεργειών, η ε, είναι επίσης κάτι το οποίο χρησιμοποιεί τα ζωτούχα λοιπάσματα με καλύτερο, πιο οικονομικό τρόπο και βελτιώνει και τη χρήση του εδάφους. Υπάρχει μεγαλύτερη ε, 15 με 25% μεγαλύτερη, καλύτερη, περισσότερη απόδοση μετά από την πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται τα λοιπάσματα. Όταν αλλάξει η καλλιέργεια δηλαδή τώρα. <clears throat> Ε, τα ευρύτερα περιβαλλοντολογικά ωφέλη για τον κύκλο του αζότου. <clears throat> Μιλήσαμε ότι χρειάζεται, είπαμε ήδη ότι χρειάζονται λιγότερα λοιπάσματα, αλλά υπάρχει και χρειάζεται και λιγότερα ορυκτά καύσιμα για να παραχθούν τα λοιπάσματα αυτά και λιγότερη εκπομπή ε, αερίων όπως το αζωτούχων αέριο όπως το μονοξίδιο του αζότου που είναι χαμηλότερες για τα πρωτεϊνούχα από ό,τι για άλλες καλλιέργειες. Άλλο σημαντικό περιβαλλοντολογικό στοιχείο είναι ότι αυξάνουν τη βιοπικιλότητα τα όσπρια και τα υπόλοιπα πρωτεϊνούχα γιατί ωφελούν και τα έντομα τα οποία κάνουν την γονιμοποίηση. Εκτός από αυτήν τη διαφοροποίηση και τη βιοπικιλότητα λοιπόν, ωφελείται και το έδαφος και το υπέδαφος. Ένα από τα θέματα για τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων αφορά το τι συμβαίνει στις περιφέρειες όπου καλλιεργούνται αυτά τα πρωτεϊνούχα. Τα εισάγουμε κυρίως από την Νότια Αμερική και εδώ στην πάνω εικόνα δεξιά βλέπουμε ότι αφού έχουν καλλιεργη, έχει καλλιεργηθεί σόγια για μερικά χρόνια παρατηρείται χειροτέρευση του εδάφους και απαιτείται αλλαγή της καλλιέργειας. Άρα η σε μεγάλη κλίμακα καλλιέργεια όγιας μπορεί να είναι αρνητική μακροπρόθεσμα στις χώρες όπου καλλιεργείται. Εδώ το, τα στοιχεία είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Δείχνουν ότι δείχνουν το πώς συγκρίνουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από προϊόντα μεταποιημένα που σχετίζονται με την κτηνοτροφία και την παραγωγή κρέατος. Συγκρίνουμε λοιπόν πάνω-πάνω ζωοτροφές από όσπρια με κρέατα που παράγονται από ζωοτροφές με σόγια ό,τι πρασινότερο βλέπετε είναι καλύτερο για το περιβάλλον και φαίνεται ότι τα όσπρια είναι καλύτερα από τη σόγια για το περιβάλλον ως προς τις ενεργειακές απαιτήσεις και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Και κάτω-κάτω βλέπουμε ότι είναι πιο οικονομική η παραγωγή ζωοτροφών επιτόπου από όσπρια. η ανάπτυξη της κατανάλωσης πουλερικών και χειρίου κρέατος είναι κάτι που στηρίζεται στις εισαγωγές πρωτεϊνούχων ζωοτροφών. Έχουμε στοιχεία εδώ από το 60 μέχρι το 2010 για την παραγωγή κρεάτων τέτοιου είδους. Κυρίως βοήου κρέατος, εκεί δεν άλλαξαν πολύ τα πράγματα, αλλά στα δύο σκοτεινότερα, δύο σκοτεινότερες παραστάσεις που αφορούν τα πουλερικά και το χείριο κρέας βλέπουμε σε σύγκριση με την εισαγωγή το, της σόγιας ότι όσο αυξάνεται η κατανάλωση αυτών των κρεάτων τόσο αυξάνεται και η εισαγωγή σόγιας. Τώρα τίθενται εδώ μερικά προβλήματα στη Γεωργία ως προς την αύξηση πρωτεϊνούχων καλλιεργιών στην Ευρώπη. Εδώ στη γραφική παράσταση βλέπετε ότι μεταξύ του 60 και του 2010 στην πάνω-πάνω γραμμή τι ισχύει για την παραγωγή σιταριού στην Ευρώπη. Είναι αριθμοί από τη Γαλλία. Ο ευρωπαϊκός σίτος έχει αυξηθεί κατά τρεις φορές περίπου κατά 300% ενώ στην κάτω γραμμή, στις κάτω γραμμές βλέπουμε την παραγωγή της σόγιας στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες και εκεί βλέπουμε ότι πρόκειται για μια επένδυση στην καλλιέργεια δημητριακών που δείχνει σαφές όφελος, συγκριτικό όφελος για την Ευρώπη. Τώρα, οι τιμές των ε, λοιπασμάτων είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία αυτά φυσικά, γιατί αυξάνεται η τιμή. Εδώ βλέπετε ότι έχουν υπάρξει και παρεμβάσεις για να αυξηθεί η παραγωγή των πρωτεϊνούχων στην Ευρώπη. Η πάνω γραμμή δείχνει πως ότι έχει μειωθεί αυτή η παραγωγή μεταξύ 60 και 2010 στην Ευρώπη. Ενώ οι κάτω γραμμές δείχνουν την παραγωγή σόγιας και μπιζελιών. Και φαίνεται ότι τελικά οι παρεμβάσεις δεν αντέστρεψαν τις τάσεις που παρατηρούνται από το 60. Τώρα θα θέλαμε να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να γίνει ως παρέμβαση για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να δούμε, να βρούμε μία ολοκληρωμένη πολιτική με πολλαπλά μέτρα αν θέλουμε να γεφυρώσουμε το πρωτεϊνικό μας έλλειμμα. Αυτή η πολιτική όμως πρέπει να είναι εξισορροπημένη και αναπτυξιακή γεωργική πολιτική, να μην υποχρεώνεται κανείς να καλλιεργήσει όσπρια. Δεν καθορίζουμε λοιπόν συγκεκριμένους στόχους για παραγωγή πρωτεϊνούχων, αλλά για μείωση των αρνητικών πρακτικών, όπως την αυξανόμενη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Μια συνολική στρατηγική δηλαδή, που να μειώνει την εισαγωγή και κατανάλωση των πρωτεϊνούχων για ζωοτροφές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους χρειάζεται δημόσια παρέμβαση και ελπίζουμε να σας έχουμε δείξει μερικούς πόσο καλύτερα είναι για τους καλλιεργητές, για την ΚΑΠ 2020 και για το περιβάλλον. Και τώρα θα θέλαμε να σας δείξουμε και άλλες επιλογές. Καταρχήν πιο αυστηρή βιοπικιλότητα στις καλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της ΚΑΠ ό,τι προτείνεται δεν πρόκειται να αλλάξει τα πράγματα ουσιαστικά. Αν θέλουμε αλλαγές τότε αντί να υποκαθιστούμε ένα δημητριακό από άλλο θα πρέπει να σκεφτούμε μέτρα που να συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές καλλιέργειες και αμύψεις πορές ή μάλλον εναλλαγές καλλιεργειών. Από την αρνητική πλευρά μπορεί να έχουμε λιγότερες ελεύθερες επιλογές. Να είναι λιγότερα δηλαδή τα ωφέλιμα καλλιεργήσιμα που μπορούμε να διαλέξουμε. Έπειτα η ταξινόμηση στα πλαίσια του πρασινίσματος και του πρώτου πυλώνα. Τα όσπρια μπορούν να είναι πιο ωφέλιμα σε σχέση με τα μέτρα που ήδη ισχύουν. Δεν θέλουμε τα όσπρια να καταλήξουν να μειώσουν, καλλιέργεια όσπριων να καταλήξουν να, μειώσει, να μειώσουν τα ωφέλη από άλλες καλλιέργειες, αλλά να χρησιμοποιηθούν περισσότερο σε περιφέρειες όπου υπάρχει πολύ εντατική καλλιέργεια. Τρίτη επιλογή. Εθελοντική πολιτική στήριξη. Χρειάζονται νέες προτάσεις. Εθελοντικά προγράμματα και εδώ τίθενται βέβαια οικονομικά και πολιτικά προβλήματα. Αν όλες οι χώρες μέλη δέχονταν τέτοια μέτρα, τότε από λιγότερο του 2% των καλλιεργησίμων γεών για πρωτεϊνούχα θα μπορούσαμε να περάσουμε σε 6%. Βέβαια πρέπει να βάλουμε ένα νότατο όριο για να δούμε τι θα μας πει και ο ΠΟΕ. Οι επιχορηγήσεις όμως πρέπει να είναι ψηλές για να δουλέψει αυτή η επιλογή. Έχουμε και άλλες τρεις επιλογές στην ΚΑΠ. Η μία είναι η προώθηση των οσπρίων μέσω προγραμμάτων του δεύτερου πυλώνα. Διαφοροποίηση των καλλιεργειών χωρίς απώλεια ελεύθερης επιλογής. Μέσω μεγαλύτερης βιοπικιλότητας. Και αυτό απαιτεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για την καλύτερη δυνατή χρήση και προστασία του περιβάλλοντος. Άλλη επιλογή να αυξηθεί η στήριξη των βιολογικών καλλιεργειών διότι φυσικά αν αυξηθεί θα αυξηθεί και η ποσότητα πρίων που θα καλλιεργούνται γιατί χρησιμοποιούν λιγότερα λιπάσματα αφού φέρνουν από μόνα τους άζωτο στο σύστημα. Χρειάζεται βέβαια κάποιο πλαίσιο για αυτή τη βιολογική καλλιέργεια για να μην χρειάζεται ο καταναλωτής να πληρώνει την ύφη. Είναι βέβαια και αυτή η ακριβή επιλογή. Και δεν αφορά μόνο τα ωφέλη των οσπρίων, αλλά και γενικότερα περιβαλλοντολογικά ωφέλη από τη βιολογική καλλιέργεια. Άλλη επιλογή μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ είναι, θα ήταν επένδυση στην έρευνα και τεχνική πρόοδος που θα μπορούσε να γίνει μέσω του ορίζοντος 2020. Ξέρουμε από άλλες χώρες ότι τα πρωτεϊνούχα μπορούν να τύχουν περισσότερης έρευνας και ανάπτυξης ας πούμε για να βελτιωθεί η παραγωγικότητά τους, η αποδοτικότητά τους. Επίσης χρειάζεται περισσότερη επιμόρφωση για τα ωφέλη στους καλλιεργητές γιατί να καλλιεργήσουν προτεραιοινούχα και πώς ωφελεί αυτό το γενικότερο αγροτικό σύστημα, γεωργικό σύστημα. Βέβαια αυτό είναι και θέμα της τροφιμικής ασφαλείας. Αυτές είναι οι έξι επιλογές που σκεφτήκαμε στα πλαίσια της ΚΑΠ. Και τώρα σύντομα επιλογές εκτός ΚΑΠ τα πρωτεϊνούχα είναι φυσικά μέρος των προγραμμάτων προστασίας των ε, αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών και εκπομπών διοξιδίου. Σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή πρωτεϊνούχων. Αν μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, θα ήταν καλό αυτό για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Δεύτερη επιλογή. Τροφιμική πολιτική γενικότερα Γνωρίζετε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα κτλ. Η φορολόγηση των λοιπασμάτων είναι επίσης μία επιλογή, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι επιπτώσεις θα ήταν διαφορετικές αναπεριφέρεια και ανακαλλιέργεια και θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε πιο εντατική παραγωγή με περισσότερη χρήση αζωτούχων. Η εξισορρόπηση των ουσιών αυτών θα ήταν κάτι θετικό, αλλά υπάρχουν εκεί προβλήματα όπως ε, πόσο ακριβώς άζωτο κατακρατείται κλπ. Και η τελική επιλογή εκτός ΚΑΠ είναι η υποστήριξη πρωτοβουλειών των παραγωγών και από πάνω και από κάτω. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οργανώσεις καλλιεργητών που θέλουν να προωθήσουν την καλλιέργεια της σόγιας. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, όπως και η μεταφορά τεχνογνασίας. Έτσι λοιπόν, ως συμπεράσματα, το έλλειμμα πρωτεΐνης που έχουμε οφείλεται σε έλλειψη ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης πρωτεϊνών, πρωτεϊνούχων. Αν αυξήσουμε την παραγωγή των πρωτεϊνούχων αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο βιώσιμης και πιο ισορροπημένης γεωργίας. Και αυτό είναι το κλειδί. Πώς να καταλήξουμε σε ένα πιο ισορροπημένο γεωργικό σύστημα. Ελπίζω να έχουμε αποδείξει ότι χρειάζονται δημόσιες παρεμβάσεις και ότι η παραγωγή καλύτερων πρωτεϊνούχων για τους γεωργούς έχει και περιβαλλοντολογικά ωφέλη ωφελεί και τον Γεωργό και το κοινό γενικότερα. Οι αλλαγές που αρχίζουμε να βλέπουμε ως προ την αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και της σόγιας θα ενθαρρύνουν νομίζουμε την παραγωγή εναλλακτικών πρωτεϊνούχων. Και καταλήγω με τις εξής ευχαριστίες. Όχι μόνο εκείνους που ανέλαβαν τη μελέτη αλλά και το Legium Features Project. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστώ την καθηγήτρια Watson και τώρα ας αρχίσουμε με τις παρεμβάσεις. Μάρτιν Όσλινγκ. Μάρτιν ναι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά του συντάκτες της μελέτης και κυρίως την κυρία Γουάσον και τον κύριο Μέρφυ ε, για την παρουσίαση. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς για τη μεταρρύθμιση της γεωργίας ε, με καθυστέρηση υποβάλλεται αυτή η μελέτη για την έκθεση για τα πρωτεϊνούχα πριν από καιρό είχα την ίδια κατεύθυνση υιοθετήσει ότι το δυναμικό κυρίως των ε, οσπρίων, το τονίζω των οσπρίων στην κοινή αγροτική πολιτική, στην νέα αναδιαμόρφωση της νέας ε, γεωργικής πολιτικής πρέπει κάπου να ενταχθεί. Για παράδειγμα, όσον αφορά την καλλιέργεια των ε, οσπρίων και όχι μόνο με την πολυμορφία. Έτσι μια τεράστια ευκαιρία την χάσαμε. Αυτό που στην κοινή αγροτική πολιτική όσον αφορά τα όσπρια ή ε, τα πρωτεϊνούχα αναφέρονται είναι στις οικολογικές εκτάσεις προτεραιότητας. Με ένα μικρό βήμα είναι αυτό, αλλά δεν επαρκεί με κανένα τρόπο. Και για να το πω απλά, πριν από δύο εβδομάδες είχα πάει στην Λατινική Αμερική, στην Αργεντινή και στην Παραγουάη. Τι είδα εκεί. Αυτά που καλλιεργούνται σε εκτάσεις ε, μονοκαλλιέργειας ε, σόγιας συσχετίζονται και με τις επιπτώσεις της δικής μας γεωργικής πολιτικής. Καλλιεργούν σόγια εκεί, στην Αργεντινή, 70% των αρρώσιμων εκτάσεων, πράγμα που δεν είναι και πολύ λογικό και σίγουρα δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να λειτουργήσει έτσι όπως ε, σήμερα γίνεται. Και αυτό εν μέρει είναι δική μας ευθύνη ότι δημιουργούμε αυτή τη μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη με τη δική μας πολιτική. Είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι ούτως ή άλλως, όχι μόνο για αυτές τις καλλιέργειες σόγιας με ακραίο τρόπο, αλλά και για το ότι αποψηλώνονται δάση για την παραγωγή βοηδών, την κτηνοτροφία στην Αργεντινή. Και όλα αυτά αφορούν και τις δικές μας πολιτικές. Αυτή η διασύνδεση πρέπει να γίνει με σαφή τρόπο, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να βρισκόμαστε σε ένα ε, μετέωρο χώρο και να ε, μην ξέρουμε πού βασιζόμαστε. Συνδέεται το ένα με το άλλο. Και σε σχέση με την Νότια Αμερική της ΗΠΑ, όταν υπάρχουν καλές συγκομιδές ε, σόγιας, όλες αυτές οι καταστάσεις δεν έχουν σχέση με την αηφορία και την βιολογική καλλιέργεια. Επίπτωση πρέπει να είναι οπωσδήποτε να προαχθούν ε, ή τα πρωτεϊνούχα στην Ευρώπη. Και πάλι καταλήγουμε εδώ στην ΚΑΠ Δηλαδή με την πρώτο, πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για τη μεταρρύθμιση. Εδώ και χρόνια αναμένουμε για την έκθεση που μας έχει υποσχεθεί να συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτεϊνούχα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ υπάρχει κάποια αμήχανη σιωπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποθέτω ότι αυτό συναρτάται με τι διμερεί εμπορικέ σχέσει που δεν θέλουν να τι διαταράξουν με τι χώρε αυτέ όταν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίε και συμβάσεις με αυτέ τι χώρε δεν θέλουν να ξεκινήσουν μια δική τους πρωτοβουλία πρωτεϊνούχων για να μην διαταραθεί η ισορροπία των πραγμάτων εμπορικά. Και έτσι τι γίνεται. Στην Ευρώπη δεν ακολουθούμε αυτή την πορεία σε πολλά σημεία όπως θα έπρεπε. Οι προτάσεις που έγιναν τώρα στις διαπραγματεύσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό σημείο Συνδεδεμένες πληρωμές ε, για την καλλιέργεια οσπρίων που πρέπει να διασφαλιστεί. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το πράγμα. Θα πρέπει να έχουμε συνδεδεμένε πληρωμέ για τα πρωτεϊνούχα και να διασφαλιστούν αυτέ. Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπή. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Στην Ευρώπη χάσαμε το δυναμικό να μπορούμε να έχουμε βελτιώσεις ε, όσον αφορά τις διασταυρώσεις όταν έχουμε 1,8% των εκτάσεων για όσπρια. Καμιά επιχείρηση δεν θα ενδιαφερθεί να ακολουθήσει μια τέτοια καλλιέργεια ε, με διασταυρώσεις. Θα που δεν αξίζει τον κόπο. Και όταν έχουμε κόστος και σε άλλους τομείς, ε, ούτως ή άλλως τα όσπρια ακολούθησαν αυτή την εξέλιξη που για τους γεωργούς θα πρέπει να πούμε ότι σωστά λένε δεν αξίζει αυτό. Πρέπει λοιπόν να ε, επενδύσουμε σε βάθος στις επενδύσεις όπως και σε σχέση με τις πρωτοβουλίες στο Δούναβι για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων αλλά να δούμε και άλλους τομείς ως πρίον, όπως ε, για παράδειγμα τα ε, Μπιζέλια, τον Αρακά, είναι δυναμικό που δεν τον εκμεταλλευόμαστε στην Ευρώπη. Οι θετικέ επιπτώσει για το περιβάλλον δεν χρειάζεται να τονιστούν και πάλι για άλλη μια φορά. Εγώ ίδιο είμαι βιοκαλλιεργητή και για τα όσπερ είναι σημαντικό αυτό και η δέσμευση του ε, αζότου ε, με την παραδοσιακή γεωργία μπορεί να είναι αυτό σε σχέση με την παραδοσιακή γεωργία ένα τεράστιο μέτρο εξοικονόμηση ε, αζωτούχων και πρέπει αυτό να συνυπολογιστεί στι προσπάθειε για τη γεωργία μας. Είμαι ευγνώμων για τις πτυχές που αναφέρθηκαν τώρα σε σχέση με αυτή τη μελέτη. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα ώστε τα όσπρια στην κοινή αγροτική πολιτική να εξακολουθούν να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την προστασία των κλιματικών αλλαγών και για την προαγωγή της βιοπικιλότητας ως κέρια σημασία σημείο και αν δεν τα καταφέρουμε με αυτή τη μεταρρύθμιση, ε, τότε τουλάχιστον στη μελλοντική αγροτική πολιτική δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε, να συνεχίσουμε να παρακάμπτουμε τη σπουδαιότητα των οσπρίων. Θα πρέπει να, να συνεχίσει να είναι ένα σημαντικό στοιχείο της μελλοντική κοινή αγροτικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Grazie, Ευχαριστώ Μάρτιν και τώρα ο λόγος στον George Λάιον. Και η Επιτροπή έχει ζητήσει τον λόγο με τον Τάσο Χανιώτη. Τζορτζ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια για την εξαιρετική παρουσίαση καθώς και την ομάδα της. Νομίζω ότι επιχορηγείται αρκετά ε, η καλλιέργεια ως πρίον στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδίως τα μπιζέλια και τα λούπινα. Ε, η μεγάλη πρόκληση ήταν ότι οι καλλιεργητές που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις επιχορηγήσεις αυτές ε, διαμαρτύρονταν για, τα, για τις φτωχές σοδιές, ιδίως όταν οι συνθήκες ε, ήταν πολύ υγρές, ε, τα φυτά σάπιζαν, έπεφταν, δεν μπορούσαν τα μηχανήματα να, τα, να κάνουν τη συγκομιδή. Και τελικά σήκωσαν τα χέρια οι γεωργοί λόγω της, μη, της έλλειψης αξιοπιστίας των καιρικών συνθήκων, ε, λόγω της υγρασίας δηλαδή. Νομίζω ότι η πραγματική πρόκληση είναι να αναπτύξουμε ποικιλίε φυτών που να μπορούν να αποδίδουν σταθερά, να έχουμε σταθερές αποδόσεις και ίσως θα μπορούσατε να εξηγήσετε για, για ποιο λόγο δεν, έχουν καταφέρει, δεν έχουμε καταφέρει γενικά να αναπτύξουμε αξιόπιστες και γερές ποικιλίε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις καλλιέργειες αυτές ε, στην Ευρώπη. Τώρα, κάτι άλλο. Παρότι οι εισοδιές αυτές είναι πηγή πρωτεϊνών, εν τέλει πάντοτε η σόγια θεωρείται η καλύτερη πρωτεΐνη για τις, ε, γαλακτο... Ε, για τις ε, θυλάζουσες αγελάδες και για την παραγωγή του γάλακτος στην κτηνοτροφία. Πάντοτε υπάρχει μια υπεροχή της σόγιας για τη χρήση της στην κτηνοτροφία. Ίσως θα μπορούσατε κάτι να μας πείτε ή να μας δώσετε κάποια συμβολή συμβουλή για να δούμε γιατί είναι τόσο σημαντική η σόγια για τα γαλακτοφόρα ζώα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, Τζόρτζ. Έχουμε και την ε, πρότασή μας για τις συνδεδεμένες ε, ενισχύσεις και θα το έχεις δει και εσύ ότι υπάρχει μια αύξηση, ζητείται μια αύξηση της καλλιέργειας πρωτεϊνούχων φυτών και υπάρχει και ένα τριμερή διάλογος που εξελίσσεται. Ο Τάσο Χανιώτη συζήτησε το λόγο και φυσικά στη συνέχεια θα ξαναδώσω τον λόγο στην καθηγήτρια Βότσον για να απαντήσει. Τάσο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τον καθορισμό κάποιων σημείων για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ επίση ε, και την κυρία που παρουσίασε και εκείνους που συνεργάστηκαν για τη σύνταξη της μελέτης ε, για την πολύ θετική σύνοψη των περιβαλλοντικών προτεραιμάτων των ε, πρωτεϊνούχων. Θα ήθελα να πω ότι όλες οι προτάσεις ε, που εντοπίστηκαν αποτελούν κατά το μάλλον ή των ε, στοιχεία υποσυζήτηση. Αυτό που είναι σημαντικό με να αποσαφηνίσουμε ευθύ εξ αρχής για αυτό το θέμα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία που συνδέονται με τους οικονομικούς υπολογισμούς του τομέα και σε σχέση και με τα περιβαλλοντικά ενδυνάμει στοιχεία. Πρέπει αυτά να μπορέσουν να συγκλίνουν. Για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε σε διαφορετική ερμηνεία των στοιχείων αυτών. Ο καλύτερος τρόπος που θα μπορούσαμε να το κάνουμε είναι να δούμε τις διαφάνειες 5 και 14. Τις διαφάνειες ε, για την εξάρτηση ε, των εκτάσεων καλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και να δούμε σε σχέση με τις ε, πολλαπλάσιες ε, καλλιέργειες ε, όσον αφορά τα δημητριακά, να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και αυτό επειδή οι πραγματικοί υπολογισμοί, και εδώ δεν έχουμε περίπλοκους υπολογισμούς, αλλά ένα σύνθετο πλαίσιο, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία, αν αντί δημητριακών παρήγαμε σόγια ή άλλα παρόμοια φυτά στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι η παγκόσμια κατάσταση που θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα δημητριακών. Η σημαντικότερη επίπτωση θα είναι χαμηλότερη παραγωγή σίτου παγκόσμια, με υψηλότερες και όλες τιμές. Και αυτό με σαφήνεια καταδεικνύει έναν οικονομικό συντελεστή που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Αυτός ο οικονομικός παράγοντας είναι που επεξηγεί γιατί σταδιακά τα πρωτεϊνούχα δεν μπόρεσαν να δραχθούν τη ευκαιρία έναντι των Δημητριακών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τι επιπτώσει. Το αντίθετο, πρέπει να μα ενδιαφέρουν οι επιπτώσει όσον αφορά τις, ε, την ένταση καλλιέργειας ε, μη ε, ε, διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων Έντονη καλλιέργεια δημητριακών. Αλλά θα πρέπει να διαρωτηθούμε περί τίνο γίνεται λόγο εδώ εναλλακτικά για τη σόγια, διότι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει οικονομικό προτέρημα, διαφορετικά θα το είχαν κάνει αυτό ήδη οι γεωργοί μα. Ή κάνουμε λόγο για τα περιβαλλοντικά προτερήματα άλλων καλλιεργειών που είναι πολύ σημαντικά. Και θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Αν όμω το πιστεύουμε αυτό, πρέπει να δούμε ποια είναι η καλύτερη μέθοδο και οδό να πετύχουμε αυτή τη σύγκληση. Πιστεύουμε ότι σωστά εντόπισαν ένα συνδυασμό πολιτικών οι ερευνητές, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα έπρεπε να μας κάνει να δούμε τις ιδιομορφίες κάθε περιοχής και κάθε χώρας για να εξεύρουμε την καλύτερη πολιτική, πολιτική προσέγγιση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα και πρέπει να το λάβουμε 100% υπόψη. Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε ότι το πρασίνισμα, η πολυμορφοποίηση, η ανακύκλωση καλλιεργιών, η αμυψισπορά είναι σημαντικά στοιχεία αλλά σε συνδυασμό, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να γεφυροποιήσουμε τα πράγματα και να διαρρήξουμε τον φαύλο κύκλο. Και θέλω να τονίσουμε ότι έχουν διπλασιαστεί τα κονδύλια σε σχέση με την έρευνα στη Γεωργία σήμερα. Και πολλά από αυτά τα κονδύλια ακριβώς θα στοχεύουν σε αυτές τις δικές μας προτεραιότητες, προσπαθώντας να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε τις καλύτερες μεθόδους για να προαχθεί η περιβαλλοντική θετικότερη επίπτωση της χρήσης αυτών των πρωτεϊνούχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή και τον Τάσο και τώρα ο λόγος ε, στον Μάρτιν. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω δύο παρατηρήσεις Πως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι θα έχουμε μείωση τη τιμή των, ε, των δημητριακών. Αλλά πώς μπορούμε έτσι σε, ένα, σε μία ήπειρο να έχουμε μόνο καλλιέργεια σόγιας όπου οι κλιματικές ε, προδιαγραφές δεν είναι τόσο διαφορετικές σε σχέση με την Ευρώπη αλλά υπάρχουν αποκλειστικά οικονομικά προτερήματα και έτσι χρησιμοποιείται η καλλιέργεια της ε, ε, σόγιας και σίγουρα αυτό έχει αρνητικότατες ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις όχι μόνο για τη γενετικά τροποποιημένη σόγια αλλά και σε σχέση, σε σχέση με τις όλες ε, συνεπακόλουθες πολιτικές. Αυτό το πρότυπο που ακολουθεί η Αργεντινή δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι αηφόρο. Υπάρχουν τεράστιες επικρίσεις. Εξαρτώμαστε από εισαγωγές από ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να διατηρηθεί Εντάξει, εμεί τι κάνουμε. Παράγουμε δημητριακά. Η Νότια Αμερική τι κάνει. Παράγουν σόγια. Είναι ένα επιμερισμό έργου, εργασία παγκόσμια, αναήπειρο, που δεν είναι σωστό. Δεν είναι αηφόρο. Και γι' αυτό δεν κατανοώ γιατί το λένε και το δέχονται. Ότι δεν υπάρχει λέει, συμφέρον για του γεωργού να ε, μειώσουν την παραγωγή δημητριακών του ε, και να καλλιεργούν περισσότερα τα όσπρια. Δεν το κατανοώ. Μία ερώτηση θα είχα προς τους συντάκτες της μελέτης. Εχθέ και πάλι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτά και θέλω κάπως στη συζήτηση αυτά να αποσαφινιστούν και να τεθούν σε ένα διάφανο πλαίσιο. Αναφερόταν για τα πρωτεϊνούχα μόνο η κράμβη. Η κράμβη δεν είναι όσπριο. Ε, παράγει παράλληλα με το έλαιο και πρωτεΐνη και χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. Εντάξει, σωστό αυτό αλλά τη συζήτηση για την Ευρώπη θα την κλείσουμε σε τόσο στενό πλαίσιο για να συζητάμε μόνο αποκλειστικά για την κράμβη. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να θέσουμε στο προσκήνιο τα όσπρια συνολικότερα λόγω των θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της καλλιεργιάς τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα δώσω τώρα το λόγο στη δόκτωρα Βότσον για να κάνει κάποια τελικά σχόλια και σας ευχαριστώ και εγώ για την εξαιρετική εργασία και για τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα που, στα οποία κατέληξε η έρευνά σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για τις ερωτήσεις να μιλήσω πρώτα για το ζήτημα της ελαιοκράμβης και μετά να περάσω στα άλλα. Οι ελαιούχοι σπόροι δίνουν λιγότερ, αποδίδουν λιγότερη πρωτεΐνη αναεκτεάρια σε σχέση με τα ψυχανθή ε, και απαιτούν και περισσότερα λιπάσματα. Τώρα, σε σχέση με κάποια άλλα θέματα για, την, για τις νέες ποικιλίε φυτών, θα ζητήσω από τον συνάδελφο τον Φρέντ Στόνταρντ να απαντήσει ως με εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας. Μάλιστα, όλα δουλεύουν, ωραία. Τα μικρόφωνα δουλεύουν δηλαδή. Η υπόθεση εργασίας ήταν ότι έχουμε αποτύχει να αναπτύξουμε νέες ποικιλίε φυτών. Ε, έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος, αλλά είναι θέμα επενδύσεων και επιστήμης και η εφαρμογή της επιστήμης στην Αυστραλία και στον Καναδά, όπου υπήρξαν πολύ περισσότερες δημόσιες επενδύσεις στις νέες ποικιλίε ψυχανθών, υπάρχει καλύτερη σταθερότητα αποδόσεων στη Σοδιά από ό,τι στις αντίστοιχες εκτάσεις της Ευρώπης. Η εφαρμογή της, επιστοσή... της επιστήμης στην Ευρώπη υπολείπεται πάρα πολύ σε σχέση με τον τομέα των σιτηρών, γιατί είναι ίσονος σημασίας. Στον κύκλο των πουλερικών και των αυγών παραμένει μικρή η συμμετοχή των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών λόγω της έλλειψης επενδύσεων και πόρων. Ωστόσο, στις διάφορες χώρες όπου έζησα, είδα ότι εκείνοι οι γεωργοί οι οποίοι προσέχουν τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, κατά κανόνα έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από εκείνους και έχω γνωρίσει παντούς που τα φυτεύουν και μετά ε, το, ξεχνούν. Λένε εντάξει αυτά τα φυτά προσδένουν από μόνα τους ε, προσλαμβάνουν από μόνα τους άζωτο και άρα δεν χρειάζεται να τα φροντίσω. Ε, οι, οι, οι γεωργοί οι οποίοι φροντίζουν Μάλλον οι γεωργοί των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών συνήθως δεν είναι πολύ καλοί γεωργοί και γι' αυτό έχουν και φτωχότερες σοδιές. Υπάρχει ένα θέμα όμως με την ανάπτυξη νέων ποικιλιών, είναι θέμα επενδύσεων. Επίσης δεν έχουμε την επιστημονική τεκμηρίωση για τα γονίδια για να μπορέσουμε να έχουμε ταχεία πρόοδο. Αυτό έρχεται όμως με την πρόοδο της γενετικής τα τελευταία χρόνια, θα τα έχουμε τα γονίδια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, η έλλειψη αξιοπιστίας και οι δυσκολίες της καλλιέργειας των καλλιεργιών αυτών, ε, είναι, τα σχετικά σχόλια ήταν πολύ εύστοχα. Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, για να απαντήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μέρφε για να απαντήσει. Θα κάνω ένα γενικό σχόλιο. Τα ερωτήματα και τα σχόλια των βουλευτών και της Επιτροπής ε, δικαιολογούνται απόλυτα από τα επιστημονικά στοιχεία, ανεξάρτητα από την άποψη που υποστηρίζει κανείς. Η συζήτηση που γίνεται εδώ είναι μια συζήτηση υψηλού επίπεδου σε σχέση με τα επιστημονικά στοιχεία. Είναι μια συζήτηση που βασίζεται σε τεκμηρίωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, έθιξε ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Η Ευρώπη είναι ένα καλό μέρος για να καλλιεργεί κανείς σιτηρά και πρωτεϊνούχα αλλά δεν έχει, είναι καλύτερη από ότι άλλες περιοχές του κόσμου. Η Ευρώπη λοιπόν έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο να χρησιμοποιεί το έδαφος της για σιτηρά και είναι μεταξύ των παραγωγών των καλύτερων σιτηρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν οι οικονομικές ε, δυνάμεις και χρειάζεται να γίνει μια ανακατανομή των πόρων προς την πλευρά των σιτηρών. Το κοινό όμως σίγουρα θα ωφεληθεί με μια καλύτερη ισορροπία. Νομίζω ότι ε, στην παραγωγή των σιτηρών έχουμε ξεπεράσει πια τα όρια. Σε μερικές χώρες ε, η εισοδιά και οι αποδόσεις των σιτηρών τελματώσει ε, και δεν εφαρμόζεται μια σωστή πολιτική άμυψης ποράς και φοβάμαι ότι στο μέλλον όχι μόνο θα έχουμε έλλειμμα ε, με τα σιτηρά αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε και την παραγωγή άλλων καλλιεργειών. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας. Σε λίγο θα εκδοθεί και η τελική εκδοχή των συμπερασμάτων της έρευνάς μας και θα μπορέσετε να τη διαβάσετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ναι, βλέπω ότι δεν θέλει κανείς να πάλι το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους. Ας περάσουμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Ωραία. Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού ε, και των συνεφών προϊόντων. Εισηγητής Ξάμπα Σάντορ Ταμπάτζη. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε στο δεύτερο στάδιο ανταλλαγής απόψεων για την προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών και διοικητικών των κρατών μελών για την κατασκευή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Είμαστε λοιπόν στο στάδιο της δεύτερης ανταλλαγής απόψεων με την Επιτροπή. Ο συνάδελφος Ξάμπα Ταμπάτζη θα μας ε, παρουσιάσει τη γνωμοδότηση και όπως είδαμε και την πρασμένη φορά, εδώ έχουμε κάποια θέματα με υψηλή πολιτική σημασία και ζητήματα υψηλώ ε, επαμφωτερίζοντα και αμφιλεγόμενα. Ε, αύριο είναι η τελευταία προθεσμία υποβολής τροπολογιών μέχρι τις 12 η ώρα 26 Απριλίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται για τις 29 και 30 Μαΐου. Τσάμπα, σου δίνω τον λόγο και ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Τσάμπα. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, με βάση τις συζητήσεις στην προηγούμενη συνάντηση αποσαφηνίζονται αρκετά θέματα και σε σχέση και με τις πτυχές όσον αφορά το περιβάλλον και τις ε, ε, δραστηριότητες της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα προαναφέρθηκαν. Ανταυτού θα ήθελα να υπογραμμίσω και να επικεντρωστώ στα θέματα τα οποία είναι πιο αμφίσιμα σε σχέση με τις θέσεις της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, στην ε, Επιτροπή Γεωργίας δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαχωριστική γραμμή όπου να υπάρχουν ιδιαίτερες τριβές. Δύο ή τρία μέλη κατέθεσαν τροπολογίες τρεις ευρωβουλευτές και προφανώς η προθεσμία είναι αύριο, είναι αύριο. Κάποια στοιχεία επί των οποίων θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή, προσοχή σας. Πρώτα, πρέπει να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων καπνοπαραγωγών σε αυτή την φάση όπου έχουμε την τροποποίηση αυτής της οδηγίας ώστε να μην διακυβευθούν τα συμφέροντά τους και να μην καταλήξουν σε μια κατάσταση η παραγωγή που να υπονομεύει τη θέση τους. Σε σχέση με τη μελέτη επιπτώσεων για την κατάσταση αυτή όσον αφορά την παραγωγή καπνού και την θέση των καπνοπαραγωγών, λέγοντας ότι δεν μπορώ να δω κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο άμεσα να ε, προδιαγράφεται εδώ, παρότι δεν υπάρχει κάποια κάποιο πρόσθετο επιχείρημα από μια μελέτη επιπτώσεων για να μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θα πρέπει να συνεχίσει να παράγεται καπνό. Σημαντικό για την Πορτογαλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία και κάποια άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει να μπορέσει να διασφαλιστεί η παραγωγή καπνού. Στο σχέδιο έκθεσής μου υποστηρίζω ότι για την δυνατότητα παραγωγής αυτής της ε, καλλιέργειας καπνού λέμε ότι θα μπορούσε στην επεξεργασία του καπνού να μπορεί να χρησιμοποιείται ε, το μπάλι, το μπάκο με την χρήση της ζάχαρης ως προσθήκης. Αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά υποστηρίζεται ευρύτερα. Είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος να ληφθεί υπόψη αυτό το σημείο. Δεν υπήρξε αμφισβήτηση ούτε χθε ούτε ε, προηγούμενα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και να διασφαλίσουμε αυτή την ε, κατεύθυνση για τους ε, Ευρωπαίους καπνοπαραγωγούς. Θα ήθελα να ζητήσω να υποστηριχθεί αυτή η πρόπτικη. Δηλαδή, κάνουμε λόγο για τη δημιουργία ενός ταμείου πρόληψης του καπνίσματος και σε σχέση με την πρόληψη του καπνίσματος είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Ταμείο Πρόληψης Καπνίσματος και όσον αφορά και τις ε, δυνατότητες ε, στο διαδίκτυο θα πρέπει να απαγορεύεται το εμπόριο ε, και οι πωλήσει μέσω διαδικτύου ηλεκτρονικά και από πλευρά του εισηγητού έχω καταθέσει και εγώ τις δικές μου προτάσεις η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος υποστηρίζουν με άλλα λόγια αυτή την προσπάθεια. Τώρα σε σχέση με την δική μας Επιτροπή ζητώ πραγματικά να υποστηρίξετε την απαγόρευση στο διαδίκτυο των πωλήσεων αυτών των προϊόντων καπνού διότι αυτό είναι ιδιαίτερα βλαπτικό για τους νέους και από την άλλη πλευρά συνεπάγεται τεράστιους κινδύνους όσον αφορά το εμπόριο παράνομων ε, προϊόντων, προϊόντων ε, απομίμησης ε, μαϊμούδων. Αν δούμε ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε και το πρόβλημα με τα τσιγάρα. Πρέπει ένα σεμινάριο να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα καπνοπαραγωγή θα υποστούν τις επιπτώσεις ε, των ε, τσιγάρων αυτών των ηλεκτρονικών τσιγάρων και πρέπει ιδιαίτερα προσεκτικά να λάβουμε υπόψη αυτή την προοπτική και να δούμε τι συμβαίνει με το εμπόριο αυτών των προϊόντων. Όπως ε, πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη το ε, τοποθετήσεις που είναι ιδιαίτερα ε, στεναρές σε αυτό. Αν δεν διαφοροποιήσουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ προϊόντων καπνού σε σχέση με τα φύλλα καπνού ως συστατικού στοιχείου του καπνού και αν δεν υπάρξει μια διαφοροποίηση όσον αφορά τις ουσίες που εμπεριέχει το, ο καπνός όσον αφορά τις συστατικές ουσίες του τότε μπορεί να καταλήξουμε με προσφυγή σε δικαστήρια και να καταλήξουμε σε ε, θέματα τα οποία θα τεθούν υπό δικαστική δικαιοδοσία. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι μόνο απλά ένα ζήτημα υποθετικών περιπτώσεων είναι ένα χειροπιαστό καθημερινό πρόβλημα που αφορά την καθημερινή ζωή. Και πρέπει εδώ με έναν αρνητικό κατάλογο, π.χ. στη Γερμανία και στο Βέλγιο, Γερμανία και Βέλγιο ως ε, παράδειγμα για την ε, ε, χρήση ουσιών που αλλοιώνουν τη γεύση, επηρεάζουν τη γεύση, γευστικές ουσίες. Σε σχέση με όλα αυτά πρέπει στην πρακτική εφαρμογή να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και από πλευράς Επιτροπής Περιβάλλοντος ο εισηγητή θεωρεί ότι η εμπορία οποιονδήποτε νέων τέτοιων τύπων σιγάρων θα πρέπει να συναρτάται με αυτό ακριβώς το ζήτημα της χρήσης για παράδειγμα τέτοιων ουσιών να μην είναι δυνατόν οι ε, καπνοβιομηχανίες να χρησιμοποιούν αδιάκριτα τέτοιου είδους γευστικές ουσίες που μπορούν να διακυβεύουν την, την υγεία ακόμα και των νέων ε, καπνιστών. Και πρέπει να δούμε εδώ σε σχέση με το Βέλγιο και τη Γερμανία αυτή την προοπτική. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ποιες γευστικές ουσίες θα επιτραπούν και ποιες θα απαγορευθούν. Και στρεφόμενοι τώρα στις ε, επιμέρους συσκευασίες αυτό σε σχέση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι ένα πολύ σημαντικό, επίμαχο θέμα. Αν δει κανείς τι συμβαίνει στην Αυστραλία και το τι συμβαίνει με τις ε, συσκευασία στην Ευρώπη, συμφωνώ με την κυρία Κλάς, δεν παρίσταται αυτή τη στιγμή, αλλά συμφωνώ με εκείνους που εκφράζουν την άποψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερρύθμιση αυτού του τομέα και υπάρχουν υπερβολικά αυστηρές διατάξεις ε, και ε, κανονισμοί. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Όταν κάνουμε λόγο για χιλιοστόμετρα στην επιφάνεια συσκευασιών. Αν δει κανείς το πακέτο των τσιγάρων, ε, θα έπρεπε να έχουμε ένα συγκεκριμένο μέγεθος για αυτές τις ε, διατάξεις. Δεν πρέπει να ε, επεμβαίνουμε σε υπερβολικό, υπερβολικά λεπτομερές επίπεδο ρύθμισης. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα εθνικό περιθώριο που θα αφήνουμε ε, για να δράσουν τα κράτη-μέλη. Εφόσον θα ενημερώνονται οι καταναλωτές ε, για το βαθμό στον οποίο τα καπνοπροϊόντα βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και είναι ιδιαίτερα βλαπτικά στην ανθρώπινη υγεία, ε, τότε η προστασία ακριβώς των καταναλωτών είναι το πιο σημαντικό ως προτεραιότητα. Να ενημερώνονται οι καταναλωτές ότι όλα τα καπνοπροϊόντα είναι επικίνδυνα και ο βαθμός τώρα επικινδυνότητας ε, είναι κάτι άλλο. Αυτό το οποίο εγώ προτείνω είναι να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος, ένα, μία μαύρη επισήμανση, ε, δύο αν είναι περισσότερο επικίνδυνο, τρεις τέτοιες μαύρες επισημάνσεις ως σήματα αν είναι άκρος επικίνδυνο. Λοιπόν, δεν υπάρχει με άλλα λόγια κάποιο ουσιαστικό επιχείρημα γιατί να μην μπορούμε να ενημερώνουμε τους ε, καταναλωτές για τους κινδύνους τους κινδύνους που συνεπάγεται το να καπνίζει κάποιος ένα σιγάρο Καλό θα ήταν εδώ αν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τίνει ευήκονους και να αφουγκραστεί τις απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Διότι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αρκετοί αγορητές ε, τοποθετήθηκαν επ' αυτού και το ίδιο συμβαίνει και εδώ και συμπερασματικά υπάρχει ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει ακόμα να αναφερθεί και κάτι το οποίο έχει υποστηριχθεί και από τους συναδέλφους είναι η εφαρμογή, η ε, υλοποίηση των κατεξουσιοδότηση πράξεων, των ε, κατεντολήν πράξεων. Η κατεξουσιοδότηση δραστηριοποίηση στη σημερινή συγκυρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αναλαμβάνει υπερβολικές εξουσίες και δεν μπορούμε κάτι τέτοιο να το δεχθούμε αδιαμαρτύρητα. Υποστηρίζουμε μια πρόταση που θα πρέπει να μας κάνει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες αυτής της κατάστασης και το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο να έχουν μια ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους επ' αυτού και να μειώσουμε τον αριθμό των κατεξουσιοδότηση πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε την άλλη εναλλακτική πορεία αν ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν πολλοί που έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριο κύριος Σπύρος Δανέλης και μετά η κυρία Λούλινγκ. Σπύρος παρακαλώ. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι ε, κεντρική υποχρέωσή μας είναι η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών και η προστασία της δημόσιας υγείας. Βέβαια, δεν μιλάμε για την απαγόρευση των καπνικών προϊόντων, αλλά μιλάμε για τη ρύθμιση της αγοράς τους. Συμφωνώ απολύτως με την κεντρική ιδέα του Ξάμπα ότι το πιο ισχυρό εργαλείο για την αποτροπή της προσέλκυσης κυρίως νέων ανθρώπων στο κάπνισμα είναι η γνώση, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση. Και με βρίσκει απολύτω σύμφωνο η πρότασή του για τη σύσταση ενός ισχυρού Ευρωπαϊκού Ταμείου πρόληψης του καπνίσματος. Νομίζω ότι η κεντρική οπτική γωνία για τη δική μας την Επιτροπή, για την Επιτροπή Γεωργίας, δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η προάσπιση των 400.000 περίπου θέσεων εργασίας για τα καπνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι μιλάμε για κοινωνικά μειονεκτούσες περιφέρειες που παράγουν καπνά στην Ευρώπη με σχεδόν μηδενικές δυνατότητες εναλλακτικής καλλιέργειας. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι τα τελευταία δύο, ίσως και τρία χρόνια υπάρχει παγκόσμια μια υποκριτική και προδήλως ύποπτη προσπάθεια αποκλεισμού των ευρωπαϊκών καπνών και υποκατάστασή τους στην αγορά από καπνά του τρίτου, των τρίτων χωρών, κυρίως τα Βιρτζίνια. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι τα, η μεγάλη πλειοψηφία των παραγόμενων στην Ευρώπη καπνών, που είναι ανατολικού τύπου και μπέρλεϊ, για να είναι εμπορεύσιμα χρειάζονται ως πρόσμικτη ουσία τη ζάχαρη. Έτσι είναι κεντρικό ζήτημα νομίζω για την Επιτροπή μας ώστε στην έκθεση να γίνεται απολύτως σαφής μία ότι η πρόσμιξη με ζάχαρη επιτρέπεται, όπως επίσης συμφωνώ απόλυτα με τον Ξάμπα ότι θα πρέπει να είναι σαφές το τι πρόσμικτες ουσίες επιτρέπονται και ποιες απαγορεύονται. Τέλος, ε, να πω ότι σε σχέση με το πακέτο, με την εμφάνιση παρότι δεν είναι κύριο ζήτημα της δικής μας της Επιτροπής, αυτό που με απασχολεί είναι ότι η, η του πακέτου και η κατά το όσο, όσο μεγαλώνει η, υποχρέωση για ενιαία εμφάνιση, τόσο α, αποστερείται το κίνητρο για διαφοροποίηση και η προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των επιμέρους προϊόντων από τις ίδιες τις εταιρείες. Έτσι, το ζητούμενό μας η μείωση δηλαδή κατά το δυνατόν της επικινδυνότητας ε, πάει περίπατο διότι καμία εταιρεία δεν θα έχει το κίνητρο ε, του να διαθέσει περισσότερα χρήματα για να παράγει καλύτερης ποιότητας προϊόντα. Ευχαριστώ. Grazie Spiros, mi permetto di unirmi al tuo intervento per sottolineare a Ciaba eh, che è molto importante che nella nostra opinione si tenga distinto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 ε, υπάρχουν τα θέματα παραγωγής καπνού και υπάρχουν και τα θέματα παραγωγής τσιγάρων, καπνικών προϊόντων που είναι δύο ξεχωριστοί τομείς. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε ως Κοινοβούλιο απέναντι στην πρόταση της Επιτροπής. Αυτό είναι θεμελιώδος. Γι' αυτό και πρέπει να προασπίσουμε την ε, εντολή μας ε, ε, διαπραγμάτευσης ε, για την κοινή γεωργική πολιτική και ακριβώς οι συνδεδεμένες ε, ενισχύσεις θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καλλιέργειας του καπνού. Όχι της παραγωγής καπνικών προϊόντων, αλλά της καλλιέργειας του καπνού. Η κυρία Λούλινγκ και στη συνέχεια Κορέα. Oui, euh, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ βρίσκω ότι πρόσφατα η Κομισιόν άρχισε να επιδεικνύει ένα ιδιαίτερο ταλέντο να κάνει προτάσεις που υποτίθεται ότι προστατεύουν την υγεία των ανθρώπων αλλά που τελικά έχουν επιπτώσεις πολύ αρνητικές και δεν προστατεύουν την υγεία. Τέτοιες προτάσεις έχουμε και μπροστά μας εδώ είναι ένα παράδειγμα προτάσεων που οδηγούν σε αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό στις χώρες μας. Εγώ πιστεύω ότι η πρόταση αυτή δεν προστατεύει την υγεία των καπνιστών αλλά απλώς ζημιώνει τις πιο μικρές καπνοβιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από... υπάρχει έτσι απώλεια πολλών θέσεων εργασίας και στη χώρα μου μόνο η εφαρμογή αυτής της πρότασης που είναι τρομερά υπερβολική εκ μέρους της Κομισιόν θα απολεστούν 600 με 700 θέσεις εργασίας. Είναι λίγες αλλά είναι μικρή η χώρα. Και πρόκειται για ανειδίκευτους εργαζόμενους κυρίως, συνήθως γυναίκες, ανήπαντες γυναίκες με παιδιά, μονοπυρηνικές οικογένειες. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Ξέρουμε ότι ακούγονται παντού κινήσεις για την παρεμπόδιση της καλλιέργειας καπνού. Σας έχω εξηγήσει πολλές φορές γιατί με εναντίον της πρότασης αυτής, γιατί υπάρχουν περιφέρειες στην Ένωση όπου παράγονται πολύ ειδικέ ποιότητες καπνού σε μικρές επιφάνειες και από όπου ζουν οι κάτοικοι ως μοναδικό πόρο στην Ελλάδα, στο βορρά, κοντά στη Βουλγαρία και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Όπως και όλοι, εγώ δεν καπνίζω, αλλά είμαι πολύ ανεκτική με τους καπνιστάς. Ξέρω ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και λέω στους φίλους μου που καπνίζουν να σταματήσουν, αλλά αν δεν σταματήσουν δεν σταματάνε. Τι θες ε, να τους κάνουμε. Πάντα θα υπάρχουν καπνιστές και καπνίστριες. Τα τσιγάρα λοιπόν, ο καπνός αυτός θα παράγεται στην Ένωση, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, θα ζουν από αυτό αγρότες ή θα εισάγουμε και κυρίως παράνομα αφήνοντας να επιβιώσουν μόνο οι πολύ μεγάλες μάρκες. Γιατί αν ακολουθήσουμε την Κομισιόν δεν θα υπάρχει πια χώρος στα πακέτα για να εμφαίνεται η μάρκα. Οι μικρές μάρκες λοιπόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ένωση δεν θα επιβιώσουν μετά από τέτοια νομοθεσία. Επίσης με ανησυχή η διατύπωση του σημείου 6 για την απαγόρευση που λέει εκεί προϊόντων με ιδιαίτερο άρωμα, δεν ξέρω πώς ακριβώς το λέει. Όλα αυτά πρέπει να τα πούμε γιατί δεν έχουν καμία σχέση με το κάπνισμα. Όσοι είναι καπνιστές θα παραμείνουν και πρέπει να αποφύγουμε τις υπερβολές όπως της Κομισιόν. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η απαγόρευση. Όπως και ο εισηγητής ανησυχώ και εγώ για τον πολλαπλασιασμό των κατεξουσιοδότησης πράξεων θα κατατέσω τροπολογίες και θέλω να προσθέσω το εξής. Ξέρω ότι δεν είναι πρώτη προτεραιότητα αλλά για το 13, το σημείο 13 δεν καταλαβαίνω γιατί τα πακέτα των τσιγάρων πρέπει να είναι κυβικά και να περιέχουν μόνο 20 τσιγάρα, μήκους, μάλμπορο ή κάμελ. Πιο κοντά τσιγάρα σε μαλακό πακέτο είναι πιο βλαπτικά από άλλα που είναι σε άλλου είδους συσκευασία. δεν καταλαβαίνω πια τίποτα. Αφήστε τις ιδιαιτερότητες και των βιομηχανιών. Όλα αυτά είναι υπερβολές και αντιπαραγωγικά, ιδιαίτερα μπροστά στην τωρινή κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και ελπίζω η γνωμοδότησή μας τελικά να είναι ισορροπημένη, θα προσπαθήσω να συμβάλλω και εγώ σε αυτό. σε ευχαριστούμε ο κύριος Κορέα. Gracias, ε, ε, Κυρία Κορέα, ευχαριστώ Πρόεδρος και όθηση η συγγήτρια του ΕΛΚ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισήγητη για την έκθεση που παρουσίασε για να υπάρξει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να διασφαλιστεί η καλλιέργεια του καπνού. Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή στο ότι πρέπει να προστατεύσουμε την χρήση σε σχέση με τις ουσίες που είναι ουσιώδους χαρακτήρα για την καπνοπαραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη ζάχαρης ως ουσίας. Όπως επισημάνθηκε επανειλημμένα, νομίζω ότι είναι αναγκαίο να διαφοροποιήσουμε με σαφήνεια μεταξύ της ανάγκης να μειωθούν οι ζημιές, οι βλάβες ε, από την, στην υγεία από την κατανάλωση καπνού περιορίζοντας, αντιμετωπίζοντας ε, το κάπνισμα σε σχέση με τους νέους και σε διαφοροποίηση με την παραγωγή αυτού του προϊόντος που είναι απόλυτα νόμιμη η παραγωγή και που εξαρτώνται από αυτήν πολλές οικογένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επιπλέον να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα σε σχέση με τη βιωσιμότητα αυτής της ε, καλλιέργειας στην Ευρώπη πράγμα το οποίο σε σχέση με την υγεία των ε, καταναλωτών δεν θα υπήρχε κάποια προστασία θα είχαμε, το, της υγείας τους θα είχαμε εισαγωγές που θα αυξανόντουσαν και ποιότητας πολύ χαμηλότερης ε, στον καπνό. Πρέπει να γίνει μια δεσμεύση πολιτική σαφής υπέρ της προστασίας ε, της καπνοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. Ως προς αυτά η έκθεση του εισηγητή νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και να τονιστεί περισσότερο. Η οδηγία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την, την υποχρέωση ε, σε σχέση με τη μελέτη επιπτώσεων που θα έχουν τις επιπτώσεις τους όσον αφορά την παραγωγή καπνού. Είναι πολύ θετική η θέση του εισηγητή κατά του να συμπεριληφθούν ε, όσον αφορά τη συμπερίληψη των φύλων ε, καπνού στην καπνοκαλλιέργεια και την αντιμετώπιση απειλών ε, πρέπει εδώ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο πλαίσιο αυτών οι υπερβολικές εξουσίες ε, που αναλαμβάνει. Έχω αμφιβολίες επίσης όσον αφορά την δυνατότητα να εισαχθεί αυτός ο θετικός ή αρνητικός ε, κατάλογος που αναφέρθηκε όσον αφορά τις συστατικές ουσίες για την παραγωγή που ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις επιπτώσεις όπως αναφέρεται στην γνωμοδότηση. Σε αυτό η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Γεωργίας πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους καλλιεργητές διασφαλίζοντας ότι με κανένα τρόπο τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν ουσίες που είναι αναγκαίες για την καπνοπαραγωγή ανεξάρτητα από την ένταση του αρώματος ή της ουσίας ε, που συνεισφέρουν στο τελικό προϊόν. Αυτή θα ήταν μια λύση πιστεύω για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα και ασφάλεια για τους καλλιεργητές. Από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στον εαυτό της όπως επανειλημμένα αναφέρθηκε εδώ υπερβολικές εξουσίες σε σχέση με την έγκριση στο μέλλον αποφάσεων που θα έχουν επιπτώσει σε αυτή την καλλιέργεια. Και γι' αυτό οι, οι τροπολογίες ε, που καταθέτω προβλέπουν μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Σε σχέση με την νομική ασφάλεια ε, όσον αφορά αυτή την οδηγία πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μεγάλο ε, αριθμό αμφίσιμων θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί να εξεύρει μια ισορροπία μεταξύ της δημόσιας υγείας, της επίπτωσης οδηγίας για την ε, απασχόληση που δημιουργείται από αυτόν τον τομέα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την αρχή της αναλογικότητας. Από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό να λάβουμε υπόψη την ανάγκη αυτή η οδηγία να μην δημιουργήσει μια αύξηση του παράνομου εμπορίου όπως αναφέρθηκε εδώ σε σχέση με, την, ε, με τα προϊόντα καπνού να μην υπάρξει αυτή η επίπτωση boomerang θα πρέπει να επιτηρήσουν την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη αυτή η οδηγία να μην οδηγήσει έμεσα σε αύξηση του άνομου του παράνομου εμπορίου και σε σχέση με τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για να καταπολεμηθεί η πώληση μη εγκεκριμένων προϊόντων, παρόλα αυτά υπάρχει μια αντίφαση στην τοποθέτηση αυτή της Επιτροπής, μια και τα μέτρα που προτείνονται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαν ακριβώς να οδηγήσουν σε αύξηση αυτών των παράτυπων πρακτικών. Είναι αναγκαίο από την άλλη πλευρά οι διατάξεις που θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σαφώς συμβατές με τις διατάξεις του ΠΟΕ, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και πιστεύω ότι κάποιες πτυχές αυτής της οδηγίας δεν θα έπρεπε να καλυφθούν από αυτή την Επιτροπή. Όμως θεωρώ σημαντικό ότι τα ε, μέτρα τα οποία το εκτελεστικό στην Ευρώπη ε, αντιμετωπίζει όσον αφορά και τη συσκευασία και διάφορα άλλα θέματα πάνε υπερβολικά μακριά. Δεν είναι απόλυτα σαφή τα τεκμήρια πώς ε, αυτά όλα συνάδουν με τις διατάξεις του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου επανέρχομαι και πάλι στις προτάσεις ε, του εισηγητή και θα ήθελα να του πω, να πω ότι δεν συμφωνώ πολύ με αυτό το σύστημα ε, σηματοδότη ε, για την, τις βλαπτικές επιπτώσεις των προϊόντων καπνού στη συσκευασία. Πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι το... αυτά τα επίπεδα, αν θεσπιστούν έτσι, για να επισημάνουμε το επίπεδο βλαβών, μπορεί να οδηγήσουν, συγγνώμη, να αναδιατυπώσω λέει η ομιλήτρια. Το να θεσπιστούν αυτά τα τρία επίπεδα όπως προτείνει ο κύριος ε, Ταμπαζή δεν θα ήταν απλό απλή υπόθεση υπό επιστημονικό πρίσμα. Η εισαγωγή τέτοιων δικτών από την άλλη την πλευρά αναφέρθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και χωρίς ε, κάποια επιτυχία όσον αφορά τις διατάξεις ε, για τη διαβάθμιση προϊόντων της τροφικής αλυσίδας. Θέλω να επιμείνω στην σπουδαιότητα την κοινωνική που έχει η καπνοκαλλιέργεια, ιδιαίτερα σε μειονεκτικές περιφέρειες, εκεί όπου παράγεται κατά 80% ο καπνός. Εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι 90% σε σχέση με τις καλλιέργειες αυτές που ε, ε, εντοπίζονται στην Εστρεμαδούρα, την δική μου εκλογική περιφέρεια, 26% της συνολικής αξίας των, ε, της γεωργικής παραγωγής. Η εναλλακτική λύση για καλλιέργειες σε αυτή την περιφέρειά μου είναι πολύ περιορισμένες και έτσι πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σπουδαιότητα αυτής της παραγωγής. Είναι σημαντικό αυτό για τις θέσεις απασχόλησης όσον αφορά τον αριθμό αναεκτάριο και όσον αφορά την προσπάθεια την ένταση εργασία σε σχέση με άλλε καλλιέργειε. Αυτό ο τομέα λοιπόν δημιουργεί πολλέ θέσει εργασία μέσα σε περιοχέ σύγκληση που κατηγοριοποιούνται σε περιοχέ σύγκληση όσον αφορά τον μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος τώρα και μετά Σκότα. Tackar ordförande och Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Νομίζω ότι γενικά έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά πρέπει να κάνω και μερικά σχόλια. Είναι νομίζω δύσκολο θέμα για συζήτηση στην χώρα μου τη Σουηδία ιδιαίτερα. Ίσως να κατανοείτε ότι πρέπει να σας πω μερικά για το ενόπνευμα αντί για την νοικοτήνη. Το ενόπνευμα είναι εξίσου βλαπτικό από την άποψη της δημόσιας υγείας με την νοικοτήνη. Ξέρουμε ότι και μικρό ποσοστό ενοπνεύματος, 2 εκατοστό λίτρα ουίσκι ή μισό ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα είναι χρήσιμο αλλά δύο ποτήρια κρασί την ημέρα δεν είναι χρήσιμα. Στην Ευρώπη όμως έχουμε μια, ένα θέμα πολιτιστικό ταυτότητας και η επίκριση του κρασί, κατανάλωση κρασιού στην Ιταλία ή τη Γαλλία θα ήταν καταστροφική από πολιτικής απόψεως, έτσι δεν είναι. Στην Ιρλανδία, τη Σκοτία και αν πούμε ότι το ουίσκι είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας δεν θα γίνονταν δεκτό πολύ εύκολα. Στη Σουηδία δεν έχουμε κρασί. Έχουμε όμως. Έχουμε όμως λέγω... Δεν έχουμε γι' αυτό πρόβλημα πολιτιστικό με το ουίσκι, αλλά έχουμε το λεγόμενο σνούς. Οι άλλοι το λένε σνάφ, άλλοι σνάψ. Το σνούζ είναι καπνός για που χρησιμοποιείται από τη μύτη. Ε, πωλείται σε σακουλάκια όπως το τσάι και είναι από τα σοβαρότερα θέματα, ήταν από τα σοβαρότερα θέματα στο δημοψήφισμα που είχαμε κάνει για την ένταξη στην Ένωση. Ένα από τα μεγάλα δηλαδή θέματα ήταν και αυτό, αυτού του καπνού τόσο σοβαρό θέμα ώστε χρειάστηκε να ζητήσουμε εξαίρεση γιατί στην Ένωση απαγορευόταν αυτός ο καπνός. Έχουμε λοιπόν εξαίρεση που μας χορηγήθηκε από τη συνθήκη ένταξης ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε αυτού του είδους τον καπνό προς μάσηση ή αποτιμήτη. Δεν τον πουλάμε όμως στις άλλες χώρες της Ένωσης. Τι έγινε λοιπόν. Τεράστια φασαρία, 85% των Σουηδών δήλωσαν ότι θα θέλουν, θέλουν να βγουν από την Ένωση αν απαγορευτεί αυτός ο καπνός. Τεράστια καμπάνια λοιπόν, ώστε να επιτρέπεται και η εξαγωγή του και αυτό πρέπει να ήταν και πολύ κερδοφόρο για τους παραγωγούς. Δεν είδα ποτέ να δαπανώνται τόσα πολλά χρήματα σε διαφήμιση και λόμπινγκ όπως η Σουηδική καπνοβιομηχανία. Και είμαι πεπισμένη ότι έχετε δει και εσείς ε, αυτές τις μπροσούρες που λένε ότι είναι πολύ χρήσιμος ο καπνός αυτός σε σύγκριση με τα τσιγάρα, πολύ ωφέλιμος. Εγώ είχα την εξή θέση. Για μένα είναι σημαντικό να επιτραπεί στη Σουηδία να διατηρήσει την εξαίρεση της αυτή, αλλά επίσης σημαντικό είναι να μην της επιτρέπεται να πωλείται στη διεθνή αγορά. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα είδη νικοτίνης, όπως δεν χρειαζόμαστε και περισσότερα είδη οι μορφές ινοπνεύματος, μαριχουάνας κλπ. Υπάρχουν ήδη αρκετές. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα χρειαστεί να κάνω τροπολογίες ή αντιπροτάσεις, αλλά επιμένω να διατηρηθεί η εξαίρεση της Σουηδίας για το σνούζ. Τώρα το τι μορφή πρέπει να έχει, τι περιεχόμενο ακριβές και τα λοιπά είναι εθνικό θέμα από εκεί και πέρα. Θέμα όχι της Κομισιόν ή της Ένωσης. Πάντως δεν το πουλάμε αυτό το καπνό στους υπόλοιπες χώρες. Και δύο πρόσθετα ακόμη θέματα. Ελπίζω να τα κατανοήσετε και αυτά. Είναι δύσκολο να επιχειρηματολογήσει κανείς για αυτό το θέμα. Πολλοί με έχουν κατηγορήσει ακόμη και για εθνικισμό. Σήμερα οι καπνοβιομηχανίες λένε ότι αν εισαχθούν νέοι κανόνες και περιορισμοί θα καταλήξουμε σε περισσότερο λαθρεμπόριο. Το λαθρεμπόριο όμως δεν έχει καμία σχέση με τη μορφή των πακέτων τσιγάρων και τι θα γράφουν αυτά επάνω. Το λαθρεμπόριο αφορά μόνο την τιμή του πακέτου. Αν δεν κερδίζει κανείς από το λαθρεμπόριο δεν θα λαθρεμπορεύεται. Δεν είναι θέμα του, της μορφής του πακέτου. Υπάρχει το θέμα της φορολόγησης, Πόσο κερδοφόρο δηλαδή είναι το λαθρεμπόριο. Και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Δεν μπορώ να αποτιμήσω ακριβώς το ποσοστό βλάβης της υγείας από τα τσιγάρα γιατί δεν είναι όλα τα τσιγάρα τα ίδια. Τζαν Κάρλο, e ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω πρέπει να υπογραμμίσουμε πόσο σημαντικό, πόσο σημαντικό είναι να πούμε πόσο επίμαχες είναι οι διατάξεις αυτές, αυτής της οδηγίας. Τόσος πολλής λόγος έχει γίνει ακόμα και ο στόχος της οδηγίας είναι επίμαχος. Και υπάρχει βέβαια και το λόμπι των καπνιστών. Πιστεύω ότι κανείς δεν είναι κατά του σκοπού της οδηγίας στο Κοινοβούλιο. Το πρόβλημα είναι πώς θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Έχουμε και τη μάχη καπνιστών μη καπνιστών, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή. Δεν πρέπει να, να ξεχνούμε καμία από τις πτυχές των καπνικών προϊόντων. Μία ενημέρωση διαπαιδαγώγησης και ενημέρωσης για τους ανηλίκους και τους νέους γενικότερα είναι πάρα πολύ σημαντική. Το νεανικό κοινό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν και ξέρω ότι δεν μπορούμε εκεί να εντάξουμε αυτή την πρόταση. Πρέπει να σκεφτούμε τις περίφημες προειδοποιήσεις πάνω στα πακέτα. Δεν νομίζω ότι με την οδηγία αυτή μπορούμε να εισαγάγουμε κάποιον διαφορετικό ε, τρόπο επικοινωνίας, ε, τροποποιώντας αυτά που κάνουμε μέχρι σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτές οι προειδοποιήσεις ε, αποτρέπουν τον κόσμο από το να καπνίσει. Νομίζω ότι η φρασεολογία που θίγει την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια των ατόμων μάλλον τα οθούν να καπνίσουν περισσότερο και καθόλου δεν τα αποτρέπουν οι φρικτές εικόνες ή η φρικτή φρασεολογία. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλα οθούν τους νέους να καπνίσουν. Ευχαριστώ Τζαν Κάρλο. Λουίς Άλντες. Λουίς Άλβες και μετά Πατράουν Άλβες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά ήδη αναφέρθηκαν για την οδηγία. Πολλά από τα πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν τα προσυπογράφω. Θα ήθελα να τονίσω όμως μια πτυχή που θεωρώ ότι είναι μια έλλειψη της οδηγίας. Είχα την ευκαιρία στον Επίτροπο Μπόργο να εξηγήσω τα πράγματα στη συνάντηση και σε σχέση με την κυρία Μακάβανη Συγήτρια. Το θέμα αυτό για την οδηγία προβλέπει να μπορούν να γίνονται χάρτινες συσκευασίες ή μαλακής, ε, μαλακού χαρτιού συσκευασίες. Ωστόσο το άρθρο 9 της οδηγίας προβλέπει για το εύρος αυτών των ε, ε, συσκευασιών 55 χιλιοστά που είναι ακριβώς το εύρος της συσκευασίας το, σε χαρτί. Ωστόσο σε ήπιο μαλακό χαρτί είναι 53 τα χιλιοστόμετρα. Πράγμα που αν διατηρήσουμε αυτές τις ε, διαστάσεις σε απόλυτα μεγέθη, όλες οι συσκευασίες σε μαλακό χαρτί, αντίθετα με το 13ο άρθρο, δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγονται. Δεν θα υπάρχει χώρος ε, για να μπορούν να τοποθετηθούν οι προειδοποιήσεις ε, για την υγεία στις συσκευασίες αυτές. Θέλω να επισημάνω το πρόβλημα αυτό για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα και άλλων συσκευασιών σε σχέση με τα 53 στολίτρα που ε, παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα. Και ο κανόνας, η πρόταση σε σχέση με το άρθρο 9 είναι απλή. Δηλαδή η επισήμανση για την υγεία πρέπει πάντα να έχει όλο το εύρος ε, της συσκευασίας, με τοπική συσκευασία. Είτε πρόκειται για μαλακό χαρτί είτε σκληρό χαρτί. Σε όλο το εύρος και το ύψος το αναγκαίο ώστε να καλύπτεται το αναγκαίο ποσοστό της συσκευασία που θέλουμε. 25% προβλέπεται τώρα και το ελάχιστο ύψος για εκείνες τις συσκευασίες ώστε η εικόνα να μπορεί τουλάχιστον να ανταποκρίνεται στο ελάχιστο επίπεδο με τοπικής απεικόνησης. Ένας κανόνας αναλογικότητας ξεπερνά όλα αυτά τα προβλήματα που αυτό το απόλυτο μέτρο εισάγει ως προβλήματα και διατηρούνται οι δυνατότητες να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την, την ε, οδηγία για να μπορεί να συνεχίσει να παράγεται αυτή η συσκευασία έτσι διότι διαφορετικά θα υπάρχει εδώ πρόβλημα όσον αφορά την ίδια τη σύνταξη της ε, οδηγίας ε, σε σχέση με τις διαστάσεις, σε σχέση με το σκληρό, τη σκληρή συσκευασία. Και για τα δύο χιλιοστά λιγότερα που έχει το, σε μαλακό χαρτί η συσκευασία, πρέπει να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα θέματα της οδηγίας ε, σε σχέση με την συσκευασία σε όλο το εύρος με τοπικής απεικόνησης αλλά επίσης ε, να μπορούν και σε 66 ε, χιλιοστόμετρα να μπορούν να ε, αντιμετωπίσουν τις προδιαγραφές όπως πρέπει. Πρέπει η αναλογικότητα του μέτρου να λαμβάνεται υπόψη, γιατί αν δεν ληφθεί αυτό υπόψη, η απουσία της αναλογικότητας δημιουργεί πρόβλημα μέσω ενός κανονισμού που επιβάλλεται σε σχέση με τους παραγωγούς. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Λου. Λουίσα. Ε, η κυρία Πατράου ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ επίσης ε, την ε, έκθεση περιεκτική και εξειδικευμένη του εισηγητή μας. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την παρέμβασή μου με εκείνο που πραγματικά γνωρίζουμε σε σχέση με αυτή την οδηγία, ότι σε έξι διαφορετικέ κοινοβουλευτικέ επιτροπέ εξετάζεται αυτή η οδηγία. Αυτό είναι σημαντική πτυχή για να ξέρουμε ποια είναι η δική μα αρμοδιότητα για αυτό το θέμα. Διότι κάθε μια από τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ πρέπει να κάνει τη δουλειά τη. Και εμεί πρέπει να κάνουμε τη δική μα δουλειά σε σχέση με τι δικέ μα αρμοδιότητε. Να επιμείνουμε με σαφήνεια στα θέματα τη γεωργία. όπω είπε ήδη ο πρόεδρο, πρέπει να επιμείνουμε στου όρου παραγωγή καπνού και στου όρου παραγωγή ευρωπαϊκού καπνού αυτό πραγματικά είναι ο χώρος στον οποίο εμείς μπορούμε να κινηθούμε ως αρμοδιότητα. Αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε και εκεί πρέπει να ασκήσουμε επαρκή πίεση ώστε οι διεκδικήσεις μας και τα αιτήματά μας να περάσουν έναντι των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών και έναντι του τελικού εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτή η πτυχή είναι σημαντική. Γιατί? Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε τη δουλειά της όπως πρέπει. Έχουμε μια οδηγία εδώ για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, όμως εμείς σαφώς γνωρίζουμε μέσω μέσω της ανάγνωσης της οδηγίας ότι ξεπερνά κατά πολύ τους στόχους ε, που θέτει ενώπιόν της. Και γι' αυτό η πρώτη πτυχή που πρέπει αμέσως να επισημάνουμε και να τονίσουμε είναι ότι δεν υλοποιεί την αρχή της αναλογικότητας. Πρέπει να απαιτήσουμε πράγματι να υλοποιηθεί, να γίνει σεβαστή αυτή η αρχή της αναλογικότητας διότι ξεπερνά κατά μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο είναι αναγκαίο στα μέτρα της πρότασης και εκείνο το οποίο μπορεί να ε, ε, αποτελεί σύσταση για την εσωτερική αγορά ξεπερνούν τις αρμοδιότητές τους και τα εισκαμμένα σε σχέση με την πρόταση. Δηλαδή δεν διασφαλίζονται με κανένα τρόπο οι αναγκαίες ε, προϋποθέσεις και οι αναγκαίοι όροι για να βελτιωθούν οι όροι λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τον τομέα του καπνού. Μια άλλη αρχή που προφανώς δεν υλοποιείται και δεν είναι σεβαστή είναι η αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη-μέλη έχουν πραγματικά προτεραιότητες εδώ όσον αφορά πολλά θέματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά του. Και χωρί καμιά αμφιβολία τα κράτη-μέλη έχουν και την δυνατότητα να γνωρίζουν ποια είναι η καλύτερη στρατηγική για αυτού του τομεί. Και ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ενιαίε ιδανικέ λύσει ή ιδανική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη-μέλη. Καλύτερα θα λειτουργήσει σε κάποιε χώρε και χειρότερα σε κάποιε άλλε. Είναι δύο αρχέ που πρέπει να επιμείνουμε να γίνονται σεβαστέ. Η αναλογικότητα και, επικυρια... και τα κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή ε, η επικουρικότητα. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση. Και σε σχέση με την διεύρυνση των εντεταλμένων πράξεων ή κατεξουσιοδότηση πράξεων είναι απόλυτα απαράδεκτο αυτό. Διότι ξεπερνά τι αρμοδιότητέ τη και μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη σήμερα ή αύριο ό,τι τη γουστάρει. Το κατατοδοκούν πιστεύοντα ότι είναι το καλύτερο για αυτόν τον τομέα. Και εμεί αν δεν συμφωνούμε, η Επιτροπή Γεωργία δεν συμφωνούμε με αυτήν την κατάσταση, με αυτέ τι προτάσει. Και έτσι στο μέλλον φοβούμαι ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο αν δεν κάνουμε κάτι. Θέλω ακόμα περισσότερο να εξειδικεύσω κάποιες άλλες πτυχέ που θεωρώ ότι έχουν τη σημασία τους και αυτές. Μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα την παράλογη θέση όσον αφορά τις διαστάσεις των πακέτων τσιγάρων πράγμα που για κάποιες περιφέρειες και ιδιαίτερα στις Αζόρες θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις Πρόκειται για 133 θέσεις απασχόλησης που θα χαθούν Μπορεί κάποιοι να πούν τι είναι 133 θέσει απασχόληση. Όμω για τι Αζόρε είναι 80% σε αυτόν τον τομέα παραγωγή αυτέ οι θέσει εργασία. Και πρέπει να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανησυχητικά επίπεδα ανεργία. Εμεί κάνουμε λόγο για μια υπερπεριφερειακή περιφέρεια που είναι σε μειονεκτική θέση. Και ήδη σήμερα σε μειονεκτικέ περιοχέ παράγεται η καπνοπαραγωγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μπορούμε να καταργήσουμε έτσι την ευρωπαϊκή ε, παραγωγή ελαφρά την καρδία Μία άλλη πτυχή, η διαφοροποίηση σε σχέση με διάφορες μάρκες. Παράλογο αυτό, σε σχέση με την Επιτροπή Γεωργίας, να πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντική η ε, ταυτοποίηση κάθε ενός του προϊόντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ασυνάφεια αυτή αντιβαίνει οπωσδήποτε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα ζητήματα πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει μια αδιαφοροποίητη κατάσταση όσον αφορά αυτά που παρουσιάζονται προς το κοινό. Η μόνη διαφορά θα είναι η τιμή. Και αν μειώνεται η τιμή θα πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση. Ε, δεν είναι η κατανάλωση που θέλουμε να αυξηθεί για να προστατεύσουμε την υγεία, υγεία. Γι' αυτό όλα αυτά είναι παράλογα. Μια τελευταία πτυχή που θα ήθελα να αναφέρω και το υπογραμμίζω αυτό είναι κάποιες πτυχές όλες αυτές από τις πολλές πτυχές που έχουν υποστεί επικρίσεις όσον αφορά αυτή την οδηγία. Εδώ η εισβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την παραγωγή διαφόρων μαρκών και των διαφόρων ουσιών. Ε, ολοκληρώνω. Θα ήθελα εδώ κάπως ε, να αναφερθώ σε αυτά τα οποία ανέφερε η κυρία Λούλιν. Κάποιοι θα συνεχίσουν να παράγουν τον καπνό. Το θέμα είναι να ξέρουμε αν θα είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι ή μήπως δεν θα είμαστε εμείς και θα είναι άλλοι. Και δώσουμε κίνητρα έτσι για να αυξηθούν οι εισαγωγές, η παραγωγή καπνού και η εισαγωγή εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα ζήτημα. Θα αυξηθεί η παγκόσμια παραγωγή και θα σκοτώσουμε εμείς τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Άλμπερτ Ντες. Στη συνέχεια η Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας. Έχουμε τον Αντρέη Ρίς μαζί μας και στη συνέχεια θα κλείσει ο Τσάμπα. Albert. Ο κύριος Ντες, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Τη συζήτηση αυτή την παρακολούθησα. Δεν είμαι καπνιστής και θα ήθελα για το θέμα του καπνού να μην ε, θεωρήσω ότι ο σε επαείων. Όμως παρακολουθώντας το θέμα του καπνού και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του, πρέπει μια παρατήρηση να κάνω αν επιτρέπετε. Εννιά χρόνια είμαι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Πιο πριν ήμουνα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Πάντα ήμουνα πεπισμένος φιλοευρωπαίος. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιε αποφάσει που λαμβάνονται στι Βρυξέλλε μα το κάνουν όλο και πιο δύσκολο το έργο μα να λέμε στου ψηφοφόρου μα ότι είμαστε φιλοευρωπαίοι. Δεν μπορεί από τι Βρυξέλλε και το Στρασβούργο να καθορίζονται όλε οι λεπτομέρειε στο ευρωπαϊκό επίπεδο και σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν. Ξεκινά αυτό με τις περιγραφές των συσκευασιών και τις διατάξεις για τις συσκευασίες. Προτού τώρα ίσως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δώσει συνέχεια σε αυτό, σε όλα τα έγγραφα τα οποία εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νομοθετικές προτάσεις, στην πρώτη σελίδα ήδη θα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον 80% της επιφάνειας να καλύπτεται. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο θα ήταν ε, ε, αποδεκτό. Επικίνδυνο φαίνεται. Περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερα καψόνια, λιγότερη ελευθερία και τι θα γίνει με τις θέσεις απασχόλησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα γράφει αυτά με τον ίδιο τρόπο όταν μας υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις, όπως οι προτάσεις για τις συσκευασίες καπνού. Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Τώρα το λόγο έχει η Επιτροπή. Διευθυντής ΡΙΣ, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ο Επίτροπος θα ήθελε να σας συγχαρεί για την εργασία σας. Όπως γνωρίζετε, για την Κομισιόν είναι πολύ σημαντική η πρόταση αυτή και πιστεύω ότι είναι σημαντική και για τους Ευρώπαιους γενικότερα. Πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζει την πρόκληση της έλξης των νέων για το κάπνισμα. Ο εισηγητής υποστηρίζει τα περισσότερα από τα προτινόμενα μέτρα από την Κομισιόν όπως και τις υποχρεωτικές μεγαλύτερες φωτογραφίες και προειδοποιήσεις μέτρα ιχνηλασιμότητας και απαγόρευση της χρήσης και υποκαταστάτων. Μερικές από τις προτάσεις του εισηγητή βέβαια ξεπερνούν τις προτάσεις μας. Ε, η μία απαγόρευση διαμεθοριακών πωλήσεων το είχαμε σκεφτεί και εμείς όταν κάναμε την αξιολόγησή μας και θα ήταν υπέρ της δημόσιας υγείας αλλά τελικά προτείνουμε υποχρεωτική καταγραφή των πολιτών και διαδικασίες επαλήθευσης της ηλικία των καταναλωτών για να μειωθεί έτσι η παράνομη πώληση και διακίνηση. Η Κομισιόν μπορεί να ακούσει όμως στοιχεία και επιχειρήματα υπέρ και της πλήρους απαγόρευσης. Το άλλο θέμα, οι προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, δεν προτείνουμε την απαγόρευσή τους. ούτε την εμπορία τους γιατί μπορεί να βοηθήσουν στην, το σταμάτημα του καπνίσματος. Ταυτόχρονα δεν θα θέλαμε να χρησιμοποιηθούν σαν θύρα για να συνηθίσουν να εθιστούν οι νέοι στην νοικοτήνη. Τα προϊόντα αυτά έχουν αυξήσει πολύ την κατανάλωσή τους τα τελευταία χρόνια και θα κάνουμε μια μελέτη για να δούμε αν έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Πολλά από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στην αγορά δεν έχουν λάβει προηγούμενη αδειοδότηση ως προς την ασφάλειά τους και δεν γνωρίζουμε αν βοηθούν στο σταμάτημα του καπνίσματος. Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τους νέους και τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει ακόμα συμπέρασμα. Εμάς ο στόχος μας είναι να σταματήσει το κάπνισμα. Και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών. Άλλοι μίλησαν για εναλλακτικά μέτρα όπως διαφορετική σήμανση των προϊόντων ή δίκτες εθισμού. Πρώτον για τη σήμανση και τη συσκευασία. Αυτά είναι σημαντικό τμήμα των προτάσεων της Κομισιόν και τα σκεφτήκαμε πολύ καιρό. Ξέρουμε από επιστημονικά στοιχεία ότι οι φωτογραφίες είναι πιο αποτελεσματικές από το απλό κείμενο καθώς και τα μεγαλύτερα στοιχεία από τα μικρότερα γράμματα δηλαδή. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι είναι θέμα καλύτερης πληροφόρησης του καταναλωτή ιδιαίτερα για στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού, μεγαλύτερες προειδοποιήσεις μπροστά και πίσω στα πακέτα και αυτά που προβλέψαμε για το μέγεθος σε αυτό οφείλονται. Δεν πιστεύουμε όμως ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι στοιχειοθετείται κατηγορία, στοιχειοθετούνται τρεις κατηγορίες για σήμανση. Όπως και για τα τσιγάρα υψηλής ή χαμηλής περιεκτικότητας σε πίσα, Φάνηκε ότι οι εικόνες μιλάνε περισσότερο από τα κείμενα για τον εθισμό. Η χρησιμοποίηση αρωμάτων όπως βανίλιας ή μέντας δυός μου δεν πρέπει να επιτρέπεται γιατί αυτό διευκολύνει τον εθισμό των νέων. Και άλλες εθιστικές ουσίες όπως βιταμίνες ή καφεΐνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα τσιγάρα. ούτε ζάχαρες που δήθεν αντικαθιστούν την απώλεια ζάχαρης που δημιουργείται από, τον από τα ανατολικά καπνά. Uh, Έχουμε κάνει δοκιμές και αν δεν υπάρχει κανένα κυρίαρχο άρωμα δεν πήραμε μέτρο. Λόγω της πολυπλοκότητας της κατασκευής των τσιγάρων θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι ο ίδιος ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η πρόταση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή καπνοβιομηχανία και στην μελέτη μας προσέξαμε ιδιαίτερα όλους τους τομείς της οικονομίας μεταξύ των οποίων και τον καπνό και θυμίζουμε ότι η υπολογιζόμενη επίπτωση της πρότασης αυτής δεν θα είναι και πολύ δραματική 2% μείωση σε 5 χρόνια της κατανάλωσης 2% 2,4 εκατομμύρια λιγότεροι καπνιστές. Τώρα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις η δυνατότητα εξουσιοδότησης που προτείνουμε σχετίζεται με την ανάπτυξη με τις εξελίξεις στην επιστήμη και την αγορά. Νομίζουμε ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να διαχειριστούμε καλύτερα την αγορά. Για τα μαλακά πακέτα δεν τα απαγορεύουμε. Όσο δε για το μέγεθος των προειδοποιήσεων, στόχος μας είναι απλώς αυτού του είδους το πακέτο που δείχνω να προωθήσουμε που είναι πολύ μικρό να απαγορευτεί μάλλον γιατί εκεί δεν μπορούμε να βάλουμε τις προειδοποιήσεις και είναι και ιδιαίτερα ελκυστικό για τους νέους και ιδίως τις νέες. Τέλος, η πρότασή μας είναι φιλόδοξη αλλά πιστεύουμε ισορροπημένη. Mm. Κάριν Κάλτενμπαχ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Είχαμε, το είχα ξεχάσει πιο πριν. Είχαμε μια σειρά παρεμβάσεων και υποθέτω οι συνάδελφοι και από την βιομηχανία συσκευασία και ε, χαρτοβιομηχανία στην Ευρώπη. Η ερώτησή μου είναι στη μελέτη επιπτώσεων υπήρξαν έρευνες πώς αυτές οι νέες προδιαγραφές για τη συσκευασία έχουν επιπτώσει στην χαρτοβιομηχανία και στη βιομηχανία συσκευασιών. Αναφέρθηκε 2% μείωση όσον αφορά την κατανάλωση τσιγάρων. Τι γίνεται με αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω από τον συνάδελφο να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Προφανώς η μελέτη του αντικτύπου εξετάζει και τις επιπτώσεις στην προμήθεια. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ε, μελέτες ε, αντικτύπου που έχει κάνει ποτέ η Επιτροπή. Έχει κάνει ξεχωριστή ανάλυση για τον κλάδο, για την βιομηχανία χαρτιού, για την ε, παραγωγή καπνού και για, τα... και για το κύκλωμα χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Όπως εξηγήθηκε, ο αντίκτυπος στους καπνοκαλλιεργητές είναι ελάχιστη, ελάχιστος. Έχουμε περίπου 8.000 αγρότες στην Ευρώπη. Οι υπόλοιποι είναι περισσότερο εποχιακοί εργαζόμενοι. Η γενική μείωση όσο αφορά ε, την καλλιέργεια είναι 13 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ε, αν το υπολογίσετε θα δείτε ότι είναι ένα πολύ μειωμένο ποσοστό του τζίρου που επηρεάζεται για την χάρτο ε, χάρτοβιομηχανία Ξέρουμε ότι 10% του γενικού τους τζίρου έχει να κάνει με τα προϊόντα του καπνού. Αυτό που έχουν προετοιμαστεί για τις προτάσεις μας, έχουν εισαγάγει όλον τον εξοπλισμό, ε, τους εκτυπωτές και τα λοιπά για τις ε, τόσο για Το πρόβλημα θα μπορούσε ίσως να παρουσιαστεί ε, για τα γενικά πακέτα, τα γενώσιμα πακέτα αλλά όσο αφορά τις, ε, τα εικονίδια και τις ε, ενδείξεις μπορεί να γίνει αυτό με ελάχιστο κόστος. Νομίζω ότι ο γενικός αντίκτυπος ε, στους καλλιεργητές καθώς και στη βιομηχανία, είναι περιορισμένος και όπως και να έχει αναλογικός. Bene, Εντάξει, ευχαριστώ. Νομίζω ότι έγινε αρκετή συζήτηση με απαντήσεις. Τσάμπα, σου ζητώ να κλείσεις αυτή τη σημαντική συζήτηση και να υπενθυμίσω σε όλους ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι αύριο, 26 Απριλίου, ενώ η ψήφιση στην Επιτροπή μας προβλέπεται για τις 29 και 30 Μαΐου. Και η τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι 11 και 12 Ιουλίου. Τσάμπα, έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση ήταν εξαιρετικά σημαντική. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σε μια σειρά παραγόντων. Ο στόχος δεν είναι να μειωθεί το κάπνισμα γενικά. Ο στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός των νέων καπνιστών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Εγώ δεν είμαι καπνιστής επίσης. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν θέλουμε να καταστήσουμε τους καπνιστές από διοπομπαίους τράγους, δεν θέλουμε να τους καλλιεργήσουμε αισθήματα ενοχής επειδή καπνίζουν. Χωρίς όμως τη συνεργασία των καπνιστών, αυτή η, αυτή η οδηγία δεν θα έχει κανέναν θετικό αντίκτυπο. Ε, πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε αυτό που πρέπει μάλλον να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να, το καταλάβουμε αυτό και να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, σε αυτό. Πρέπει να θεωρήσουμε τους καπνιστές ως συμμάχους ε, στην προσπάθειά μας να πείσουμε τον κόσμο να κόψει το κάπνισμα. Θέλουμε, όπως είπα, να μειώσουμε τον αριθμό των νέων ατόμων που ξεκινούν το κάπνισμα. νομίζω ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του κυρίου Ντεκάστρο, της ε, Επιτροπής και πολλών συναδέλφων οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να γίνεται μια διάκριση μεταξύ της καλλιέργειας του καπνού και της επεξεργασίας της βιομηχανίας. Υπάρχουν 300.000 θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε και ο Σπύρος, που διακυβεύονται. Δεν δόθηκε απάντηση. Θα καλούσα την Επιτροπή να μας απαντήσει. Ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος στις εισαγωγές καπνών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν έχουμε απτά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έδωσε στοιχεία Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτής της οδηγίας ε, σε ποιο βαθμό θα δούμε μια μείωση ε, στην παραγωγή καπνού και σε ποιο βαθμό θα αυξηθούν οι εισαγωγές καπνού από άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και τώρα έρχομαι στην επεξεργασία καπνικών προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά υπάρχει και η προστασία των καταναλωτών δεν έλαβα μια ουσιαστική απάντηση από την Κομισιόν. Επιμένω πάνω σε αυτό. Επιμένουμε στο σύστημα των ενδείξεων. Αν μπορείτε να σκεφτείτε κάτι καλύτερο, μια καλύτερη πρόταση, ένα καλύτερο πλαίσιο ενημέρωσης των καταναλωτών, να σας ακούσω πολύ ευχαρίστως. Αλλά Πολλοί είπαν ότι απορρίπτουν αυτό το σύστημα επισήμανσης και ενδείξεων και προειδοποιήσεων, αλλά στις τροπολογίες δεν προτάθηκε κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα εγγυηθούμε την προστασία των καταναλωτών Αναμφίβολα πρέπει να ενημερωθούν οι καταναλωτές για κάθε μεμονωμένο προϊόν. Μιλούμε για τα ελαφρά τσιγάρα. Αν εγκαταλείψουμε τον όρο της χρήσης ελαφρών τσιγάρων, πώς θα κατανοούν οι καταναλωτές ότι πρόκειται για διαφορετικά προϊόντα. Από αυτή την άποψη θα σας ζητήσω να σκεφτείτε λίγο την καλύτερη λύση. Είναι εύκολο να πει κανείς ε, ε, πρέπει να λύσω ένα πρόβλημα, αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς πώς θα λύσει το πρόβλημα. Τώρα η αρνητική κίνδυνη σε σχέση με τα ενισχυτικά γεύσεις. Πρέπει να απαγορεύσουμε τις βιταμίνες, τον καφέ, τη βανίλια και όλα εκείνα τα προϊόντα που καθιστούν τα προϊόντα αυτά ελκυστικά για τους νέους. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια σαφή κατάσταση και στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Μάλλον υπάρχει ένα σύστημα στο Βέλγιο και στη Γερμανία γι' αυτό και μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα και η μέντα είναι επιβλαβές προϊόν. Νομίζω ότι και αυτή πρέπει να καταργηθεί ως ενισχυτικό γεύσης ή αρώματος. Συμφωνώ με την κυρία Λούλιν και τον κύριο Ντες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έχει απαντήσει. Δεν μας έχει πει ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είμαι πεπισμένος ότι αν πρόκειται να έχουμε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση και σύστημα σε σχέση με τις συσκευασίε των πακέτων, ο συνάδελφος Άλβαρες μίλησε πάνω σε αυτό και συμφωνώ μαζί του, τότε δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολική κανονιστική ρύθμιση. Συμφωνώ ότι ε, αν έχουμε υπερβολική ρύθμιση, τότε ε, χάνει την αξιοπιστία της ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν θέλω να, να προκαλέσω προβλήματα ούτε στι Αζόρες, ούτε στο Λουξεμβούργο, ούτε στην Πορτογαλία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε μια λύση που θα επιτρέψει τα μεμονωμένα πακέτα των τσιγάρων να έχουν ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη μορφή, αλλά να αφήσουμε και κάποιο περιθώριο και στην επικουρικότητα. Η ρύθμιση κανονιστική ε, δεν ε, δεν πρέπει να καταλήγει στην απαγόρευση των προϊόντων. Χαίρομαι που είσαστε υπέρ της προστασίας ε, της υγείας των ανθρώπων, ε, κυρία Αντιπρόεδρε. Φυσικά δεν πρέπει να δημιουργούμε νέες μορφές καπνού ή αλκοόλ ή ναρκωτικών, συμφωνώ. Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε όμως την σουηδική εθνική ταυτότητα και το σνούς. Υπάρχουν ε, και ιατρικές μελέτες ε, και έχει τεκμηριωθεί ότι υπάρχουν μικρότερα ποσοστά καρκίνων του πνεύματος με το σνούς. Υπάρχει αυτή η σουηδική ιδιαιτερότητα, εντάξει, να το σεβαστούμε. Υπάρχει η εξαίρεση, πρέπει να παραμείνει, γιατί είναι κομμάτι της σουηδικής ταυτότητας και δεν δημιουργεί κίνδυνο για τα άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει να το αφήσουμε στη Σουηδία πώς θα το αντιμετωπίσει. Σέβομαι τις ε, εθνικές παραδόσεις του κάθε κράτους μέλους. Μιλήσαμε για το λαθρεμπόδιο. Θέλω να περάσω το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν επιδιώκουμε μια απαγόρευση ε, των πωλήσεων των καπνικών προϊόντων. οι νέοι αγοράζουν πράγματα και μέσα από το ίντερνετ. Μπορούν να τα βρουν. Ο γενικός στόχος είναι να μειώσουμε τον αριθμό των νέων που αρχίζουν το κάπνισμα. Και αυτός είναι ο σκοπός αυτής της οδηγίας. Να απαγορεύσουμε τις πωλήσει μέσω του διαδικτύου ε, ε, είναι ένα μικρό κομμάτι, το, κομμάτι των συνολικών πωλήσεων καπνού, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να δίνουμε περιθώριο για λαθρεμπόριο ή παράνομη διακίνηση τσιγάρων και καπνικών προϊόντων. Αλλά για χάρη της προστασίας της νεολαίας πρέπει να απαγορευτεί η πώληση μέσω του διαδικτύου για τη συσκευασία τώρα. Όπως είπα και νωρίτερα για τα μεμονωμένα πακέτα πρέπει να έχουμε μια ευέλικτη προσέγγιση, μια κοινή προσέγγιση, ε, κοινή και ευέλικτη. Όσο με αφορά ας υπάρχει και εικόνα, γιατί ασκεί ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να διακυβευθούν θέσεις εργασίας και ιδίως πολλές θέσεις εργασίας. Θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ξέρετε, έχουμε την Επιτροπή Γεωργίας και είναι η, Επιτροπή των Ειδικών για τα θέματα αυτά. Εκεί που νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να προασπίσουμε τους καπνοκαλλιεργητές και ότι δεν μπορούμε να το εκφράσουμε ρητά αυτό, ότι δεν μπορού, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται η ζάχαρη, γιατί είναι ασύλληπτο είναι, είναι αδύνατο να υπάρξει παραγωγή καπνού χωρίς την προσθήκη ζάχαρης. Θέλω λοιπόν να αλλάξει η Επιτροπή αυτών των κανόνα. Πρέπει να δούμε την προστασία των καταναλωτών, τα πρόσθετα και να αποφασίσουμε τι πρέπει να απαγορευτεί και τι πρέπει να επιτραπεί. Βασικά αυτή είναι η σύνοψή μου κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ζητήσω τους συναδέλφους από το ΕΛΚ να σκεφτούν πολύ καλά κατά πόσο θα μπορούσαμε να μιμηθούμε το παράδειγμα της ε, Γερμανίας και του Βελγίου και αν κάποιος μπορεί να σκεφτεί κάτι καλότερο για την προστασία των καταναλωτών, εγώ θα αποσύρω ε, τις τρεις αυτές διαβαθμίσεις. Δηλαδή τα ελαφρά, μεσαίως ελαφρά ή δεν ξέρω εγώ. Ε, πάντως πρέπει να υπάρξει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Προσμένω τις τροπολογίες. Ε, εάν βγάλουμε μια καλή γνωμοδότηση, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προστατέψουμε και τα συμφέροντα των καπνοκαλλιεργητών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ξάμπα. Πολύ καλή δουλειά. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εύχομαι σε όλους... Ε, ε, έχουμε τελειώσει με τις εργασίες της Επιτροπής μας. Εύχομαι καλή επάνωδο για την 1η Μαΐου. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 6 Μαΐου. Ε, κυρίσω το πέρα της συνεδρίασης.